Translation is correct. Έχετε μετάφραση, ρωτάει ο Πρόεδρος. Should be okay. I think it's okay, yes. Otwieram popołudniowe posiedzenie podkomisji praw człowieka. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι να αρχίζουμε την απογευματινή μα συνεδρίαση τη Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και καλωσορίζω τον κύριο Ματσέη Ποπόφσκι που είναι αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Θα μα παρουσιάσει την επανεξέταση τη πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία. Θα μα παρουσιάσει επίση και τι πρόοδου που έχουν επιτευχθεί στον τομέα αυτό. Καλώ ήρθατε, λοιπόν. Είναι η δεύτερη φορά που σας έχουμε εδώ μαζί μας. Και διαπιστώνω ότι σήμερα θα μας παρουσιάσετε ό,τι πληροφορίες έχετε για το ταμείο αυτό, για το μέσο αυτό μετά, μπορούν να μιλήσουν και ευρωβουλευτέ, αλλά να ξέρετε ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Οπότε η πραγματική συζήτηση, συζήτηση σε βάθο θα γίνει όταν θα έχουμε εδώ την ε, το εκπρόσωπο, την ίδια την κυρία Κάθριν Άστον, το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Στις 27 Νοεμβρίου συναντηθήκαμε με την κυρία Βερονίκα Αρνό, από το Γραφείο Εκδημοκρατισμού και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία παρουσίασε στο διευρυμένο Προεδρείο μας την διάμεση εκδοχή, το έγγραφο εργασία δηλαδή, όσον αφορά τη δημιουργία του ταμείου αυτού. Επίσης, πήραμε και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα κύρια σημεία θα παρουσιαστούν το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια. Η ύπατος εκπρόσωπος, η κυρία Άστον, θα πάρει το ανακοινωθέν αυτό και θα συζητήσει με τις χώρες μέλη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια θα έχουμε σε βάθος συζήτηση εδώ στην υποπιτροπή μας μετά από την έκθεση αυτή η συζήτηση θα γίνει στις αρχές του 2012. Έχει ήδη σκιαγραφηθεί το χρονοδιάγραμμα ήδη από την προηγούμενη συνεδρίασή μας. Αυτό που θέλουμε σήμερα να ξέρουμε από εσά είναι πως έχει σήμερα η κατάσταση. Δηλαδή, ποιο είναι το αποτέλεσμα από τις διαβουλεύσεις που έλαβαν μέχρι τώρα χώρα και πώς προβλέπεται η συνέχεια των εργασιών. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της 27ης Νοεμβρίου πάντως, η πρόεδρός μας, η κυρία Μπάρμπαρα Μίλερ και λαμβάνοντας υπόψη και την άποψη του κύριου Χόβιτ, που είναι ο εισηγητής μας, έστειλαν επιστολή στην κυρία Άστον. Εκεί εξηγούν και προτείνουν πράγματα. Προτείνω πράγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ θα αναφερθώ σε ένα τμήμα της επιστολής αυτής, διότι πρόκειται για πολύ σημαντικές πληροφορίες για την συνεδρίασή μας. Η επιστολή αυτή εννοείται ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αντικαθιστά τις διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι. Αποτελεί μόνο ένα στοιχείο της προπαρασκευαστικής δουλειάς. Τα μέλη λοιπόν της υποεπιτροπής μας επιθυμούν να ζητήσουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που υπάρχουν όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων, ο κύριος Σικόσκι, Στην ομιλία του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι είναι πεπισμένος ότι μια πολιτική συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο Δεκέμβριο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας, μπορούμε να είμαστε κι εμείς εξίσου αισιόδοξοι. Οι ελπίδες αυτές του κύριου Σικόρσκι είναι βάσιμες. Θέλουμε επίσης να ξέρουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα προκειμένου να καθιδρυθεί το Ταμείο αυτό. Έχετε το λόγο παρακαλώ για να μας παρουσιάσετε το μέσο αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ποπόφσκι που με προσκαλέσατε να έρθω στην συνεδρία σε αυτή της Υποπιτροπής σας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επιτρέψτε μου να μιλήσω όμως αγγλικά, λέει ο κύριος Ποπόφσκι, μια από όλα τα έγγραφα που έχω στη διάθεσή μου και ξέρω ότι έχετε εξαίρετους διερμηνείς οι οποίοι θα βοηθήσουν στη μετάφραση. Συνεχίζει αγγλικά ο κύριος Ποπόφσκι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα αυτή που μου δίνετε να έρθω εδώ, να σας ενημερώσω για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία όπως γνωρίζετε, αλλά η ύπατος εκπρόσωπος όπως έχει προγραμματιστεί θα σας παρουσιάσει το Δεκέμβριο τις ιδέες της στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Την ε, μελλοντική στρατηγική δηλαδή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και δίχως άλλο προσδοκά και εκείνη να έχει μια καρποφόρα συζήτηση μαζί σας το Δεκέμβριο, 15 Δεκεμβρίου. Όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ το υπόβαθρο. Πέρασαμε χρόνο προετοιμάζοντας την πρόταση και τη συζήτηση και ήταν ε, απαραίτητο κατά το χρονικό αυτό διάστημα να ακούσουμε και όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι ευρωβουλευτές επίσης συμμετείχαν από την αρχή στη διαδικασία. Για παράδειγμα, όταν ε, ο προηγούμενος ε, πρόεδρος τον Ιούλιο του 2010 ε, συζήτησε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τότε είχαμε προτάσεις προκειμένου να συμπεριληφθούν στην έκθεσή μας. Στη συνέχεια έγιναν διάφορες άτυπες, άτυπες συνεδριάσεις με ευρωβουλευτές, ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες. Θα αναφερθώ σε μία τέτοια. Πήραμε επιστολές και από την κυρία Λοκμπίλερ και από τον Αντιπρόεδρο Μακμίλαν Σκοτ που βοήθησαν πάρα πολύ να προχωρήσει η διαδικασία. Είπατε εκπρόσωπος, ελπίζει να μπορέσει επίσημα να σας παρουσιάσει τις δικές της ιδέες όσον αφορά την αναθεώρηση της πολιτικής μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήδη από τις 8 Δεκεμβρίου. Πριν δηλαδή από την Ολομέλεια με ευρεία συζήτηση έτσι όπως αποφασίστηκε από τη διάσκεψη των Πρόεδρων. Στο σχέδιο, στο πρόχειρο, ε, φροντίζουμε να συμπεριληφθούν διάφορα σημαντικά σημεία τα οποία εσείς εντοπίσατε στις ανταλλαγές ε, απόψεων που είχαμε μεταξύ μας. Για παράδειγμα, να υπάρχει σαφή ισορρολογία όσον αφορά τον οικονομικό, τον οικουμενικό χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης ε, να διατυπώνεται σαφώς ποιος είναι ο ρόλος των χωρών μελών. Θέλουμε επίσης να υπογραμμίσουμε τον εξέχοντα ρόλο που έχει η κοινωνία των πολιτών και να υποβάλουμε ιδιαίτερα μέτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς αυτά λαμβάνονται υπόψη στις υπηρεσίες πρόσληψης προσωπικού. Νομίζω ότι και εσείς το έχετε υπογραμμίσει αυτό το σημείο ξανά και ξανά, ότι δηλαδή οι δικοί μας οι διπλωμάτες πρέπει να είναι καταρτισμένοι καλύτερα εκείνοι οι οποίοι απασχολούνται στη συνέχεια στις διάφορες διπλωματικές υπηρεσίες μας. Όλα αυτά τα θέματα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, δεν αντικαθιστούν βέβαια την ε, πλήρη διαβούλευση που έχουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεπώς, περιμένουμε και τη δικιά σας έκθεση του κύριου Χόβετ πρώτα απ' όλα για την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και τις σχετικές πολιτικές και στη συνέχεια την έκθεση αυτή καθεαυτή ε, σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη και την κοινωνία των πολιτών να πούνε την άποψή τους. Έγιναν συζητήσεις στο Συμβούλιο την Άνοιξη και στην ε, ε, Πολιτική Επιτροπή Ασφάλειας και τον Μάιο και είχαμε και δύο γύρους συζητήσεις στην Επιτροπή Πολιτικής Ασφάλειας και σε μια άλλη ομάδα εργασίας με διάφορες πιστολές που πήραμε από διαφορούς υπουργούς. Η κοινωνία των πολιτών επίσης έκανε πολλές προτάσεις, πολύ αξιόλογες. Είχαμε ε, συστάσεις πρώτα απ' όλα από το Φόρουμ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του 2010. Επίσης από διάφορες άλλες ε, ε, επιτροπές, ομάδες, οργανώσεις και περιμένουμε το νέο φόρουμ των μη κυβερνητικών οργανώσεων που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, αν δεν απατώμε. Τέλος, συνεχίζονται συζητήσεις και με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διάφορους τομείς πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, εσωτερικών ε, θεμάτων, δικαιοσύνης, έτσι ώστε η πολιτική μας να ευθυγραμμίζεται αυτή η διαδικασία διαβούλευση θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο μετά από τη συζήτηση που θα γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο. Περιμένουμε λοιπόν τις συζητήσεις αυτές. Τώρα, η κυρία Άστον, απατώντα στην επιστολή που έστειλαν από κοινού η κυρία Λόκμπιλερ και ο πρόεδρο τη Επιτροπή ΑΦΕΔ, ο Αλμπερτίνη, η ύπατη εκπρόσωπο δεσμεύτηκε να παρουσιάσει τι ιδέε της το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν όσον αφορά τη διαδικασία αυτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα, για το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία. Έχουμε ήδη διανύσει ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου και προτείναμε ότι είχαμε να προτείνουμε στα κράτη-μέλη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί ακόμα να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Αυτού Μέσου για τη Δημοκρατία ακόμα φέτο. Θα το δούμε στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεν το ξέρω ακόμα με σιγουριά γιατί τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να έχουν κάποιες ερωτήσεις. Τίποτα το φοβερό όμως. Έτσι κι δημιουργούμε κάτι καινούριο, άρα χρειάζεται χρόνος για να το προετοιμάσουμε καλά. Η βασική ιδέα όμως είναι ότι θα συνεχίσουμε και του χρόνου και θα θέλαμε να ξεκινήσει στα μέσα του 2012. Ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αυτό θα το συζητήσει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και θα υποβάλει συστάσεις προς το Συμβούλιο. Εμείς έχουμε επαφές με τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές και ευχαρίστως να λάβουμε υπόψη μας τις παρατηρήσεις σας και τις επικριτικές. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ε, κονδυλίων, τα οποία δεσμεύονται εδώ. Αυτό που ακόμα κοιτάμε και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε από κοινού να προτείνουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Αυτό είναι να δημιουργηθεί σαν καταπίστευμα, έτσι ώστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να μπορούν από κοινού να συνεισφέρουν με κονδύλια. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ελεκτική δομή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη θα εκπροσωπούνται και θα υπάρχει κάποιος πολιτικός έλεγχος για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μέσο αυτό. Δεν πρόκειται για ένα εντελώ νέο. Δεν χρειάζεται ένα καινούριο, ένας καινούριος θεσμός. Θα είναι ένα ίδρυμα που θα εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εντολή θα επικεντρωθεί στην δράση στήριξης δράσεων για τη δημοκρατία. Δημοκρατία ε, στα πλαίσια της γειτονίας μας, ανατολικά και δυτικά. Συνεπώς, το μέσο αυτό δεν θα είναι έτοιμο στα τέλη της χρονιάς, αλλά η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαύσκη. Στις 8 Δεκεμβρίου η Επιτροπή ΑΦΕΤ θα κάνει μια συζήτηση για την έκθεση αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να προωθήσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Χάουετ έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Καλωσορίζω την παρουσία του κυρίου Ποπόφσκη εδώ. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις ε, εσωτερικά για το τι θα κάνουμε στο Κοινοβούλιο για την έκθεση αυτή και μεταξύ μα έχουμε συζητήσει και με τους συναδέλφους και με τους υπολείπους ε, ε, στην Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων και πρέπει να πω ότι η έλλειψη σαφήνειας για το πώς θα ξεκινήσει και θα δεξαχθεί όλη αυτή η διαδικασία αποτελεί δυσκολία. βάση περιπτώσει είμαστε εδώ που είμαστε. Η κινητοποίηση για να υπάρξει μια μη γραφειοκρατική διαδικασία που θα βασίζεται στο διάλογο με τις ε, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί ένα πολύ καλό κίνητρο, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να τονίσουμε ότι υπάρχει έλλειψη σαφήνειας που δεν μας έχει διευκολύνει καθόλου τη ζωή. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο πέραν αυτού και ε, βεβαίως θα αποσταλούν ε, μέσω της Προέδρου και προσκλήσεις σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες για να συζητηθεί το θέμα αυτό. Όλοι θα παρέμβουμε. Θα δείτε και εσείς ποια είναι λοιπόν η θέση μας. Θα δούμε τι θα γίνει και στην Ολομέλεια του Δεκέμβρη. Λυπούμε που Μέχρι τώρα η συζήτηση έχει επικεντρωθεί στα διαδικαστικά και όχι στα ουσιαστικά της υπόθεσης. Ε, ας είμαστε ειλικρινείς. Έτσι είναι το πράγμα δυστυχώς. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει κέντρο βάρους η συζήτηση και να περάσουμε στην ουσία, γιατί δεν θα υπάρξει, δεν κάνουμε συχνά αναθεώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε αυτό είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία που έχουμε για το πώ προωθεί και σέβεται τον, την νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα η Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνώ. Ας μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Πρέπει να συζητήσουμε όλε αυτές τις διαδικασίες, ναι, αλλά ας μπούμε και στη λεπτομέρεια τελικά και στην ουσία του κειμένου που θα υποβληθεί. Να πω επίσης για, για την επιστολή που έστειλε η κυρία Λοχμπίλερ Ευχαριστώ που αναφερθήκατε και στη δική μου έκθεση, γιατί η πρόθεσή μας τελικά, μέσω αυτή τη έκθεση. ήταν να βοηθήσουμε το Κοινοβούλιο να συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία, εφόσον βεβαίω υπάρχει επίσημη επικοινωνία για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια έκθεση μεταγενέστερα. Για, την, για, τους, για την εκπρόσωπο ξέρω ότι δεν θέλει να υπάρξει διάδοση υπό των εκπροσώπων η κυρία Άστον. Αν υπάρχει ένας ύπατος εκπρόσωπος ε, ουσιαστικά ε, τραβάει τα φώτα πάνω του και δεν φαίνεται τόσο πολύ η δουλειά που κάνει η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Ε, το ερώτημα όμως είναι τι κάνουμε με τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει για τους διάφορους τομείς πολιτικής. Εγώ λοιπόν έχω πιστεί ότι το να υπάρχει ένας ύπατος εκπρόσωπος που θα συμβουλεύει την ε, Βαρονιά για θέματα διεθνούς δικαιοσύνης είναι σημαντικό. Οι Αμερικανοί το έχουν, εκπροσωπούνται παντού σε ό,τι αφορά το Διεθνές Παιδικό Δικαστήριο, ας πούμε, παρόλο που δεν είναι συμβα... ε, συμβαλόμενο μέρος. Οπότε νομίζω ότι θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για μια τέτοια θέση. Επίσης, εδώ στο Κοινοβούλιο θα θέλαμε μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας και για το, για το ρόλο που έχει να παίξει το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό όλες αυτές οι συζητήσεις που γίνονται εμπιστευτικά για να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση όταν, υπάρχει, όταν υπάρχουν περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά υπάρχουν και ευθύνε έτσι ώστε να υπάρχει λογοδοσία και για τις δικές μας δράσεις. Και νομίζω ότι αυτό δεν φαίνεται τόσο πολύ στο κείμενο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κάτι γι' αυτό. Μετά, για το διάλογο που υπάρχει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι αυτοί οι διάλογοι ε, είναι σημαντικοί μεν, αλλά δεν ε, έχουν ως κεντρικό τους θέμα ας πούμε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν ε, είναι αποτελεσματικοί, έχουμε δει διάφορες εξολογήσεις, έχουν υπάρξει αρκετά επικριτικά σχόλια. Οπότε πρέπει να δούμε ποιος είναι τελικά ο ρόλος όλας αυτής της διαδικασίας διαλόγου. Και αυτό δεν φαίνεται επαρκώς στο κείμενο. Επίσης, αναφέρθηκε ο κύριος Ποποφσκή ήδη στην ενίσχυση της διατύπωσης για το ρόλο των κρατών μελών. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει και νομίζω ότι το λέει και καλόπιστα. Αλλά αυτό που ψάχνει το Κοινοβούλιο, αυτό που ζητά και το Κοινοβούλιο και άλλοι, είναι ο μηχανισμός. Αν πούμε ότι εμείς ως κρατημέλη συμβόμαστε απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα και επομένω μπορούμε να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που τελικά θα το κάνουμε αυτό. Ποιος είναι, πού είναι ο διάλογος ο διαδραστικός που, και πού συμβαίνει. Γιατί προς το παρόν δεν λέει κάτι το κείμενο ως προς αυτό. Και έχω τη συνάδελφο εδώ την κυρία Γκόμες δίπλα μου και έχουν υπάρξει και άλλοι συνάδελφοι που εμπλάκησαν στη συζήτηση για τα χρηματοδοτικά μέσα. Και ήταν πραγματικά πολύ καυτή αυτή η συζήτηση. Έχουμε σαφείς δεσμεύσεις και από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν σε σχέση με το τι θα γίνει για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για, τα, για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μετά το 2014 όπου θα υπάρξει δηλαδή ένα επίπεδο λογοδοσίας και από την δική μας πλευρά θα υπάρξει και δυνατότητα ελέγχου. Ελπίζω η ανακοίνωση τον Δεκέμβριο να αντικατοπτρίζει και να παρουσιάζει αυτές τις δεσμεύσεις που έχουν υπάρξει ήδη, έτσι ώστε να έχουμε μια σαφή συγκεκριμένη δέσμευση σε σχέση με το μέλλον. Δεν θα μπω ε, σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά εγώ πραγματικά είμαι πολύ αισιόδοξο για το ε, ε, μέσο αυτό. Βεβαίω πρέπει να υπάρξει και επαρκή έλεγχο του προπολογισμού ω προ αυτό, αλλά πρέπει να δούμε και τι κάνουν και οι Αμερικανοί και τι κάνουμε εμεί. Νομίζω ότι έχουμε μείνει πίσω. Α μην υπάρξουν επικαλύψει. Αλλά νομίζω ότι και ένα από τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε από την Αραβική Άνοιξη είναι ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περισσότερο γίνεται για να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελπίζω να έχετε την πολιτική θέληση, να το παρακολουθήσετε, να το προωθήσετε και εμείς ε, ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο να σα υποστηρίξουμε όσο δυνατόν περισσότερο για την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες. Χωρί μικρόφωνο, κύριε Γκόμε. Για τα προπαρασκευαστικά. Αυτή η νέα στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή θα κάνει μια διαφορά. Δεν θα είναι κάτι το συνηθισμένο. Και νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι προκύψει θα είναι αποτέλεσμα ουσιαστικών διαβουλεύσεων με την κοινωνία των πολιτών και με το Κοινοβούλιο βέβαια. Υπάρχει έκθεση του Ρίτσαρντ σχετικά με το τι έχει γίνει, αλλά υπάρχει και μια προσέγγιση για το, σχετικά με το μέλλον και ποια είναι η συμβολή προς την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα ήταν μήπως καλύτερο στην Ολομέλεια του Δεκέμβρη η Λέδη Άστον να μας δώσει το δικό της όραμα, τη δική της άποψη και να συνεχίσουμε την ε, όλη διαδικασία διαβούλευσης, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να αλλάξουν. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε σαφώς ότι δεν μιλούμε απλώς για αρχές και αξίες, μιλούμε για υποχρεώσεις, νομικές υποχρεώσεις, διεθνείς νομικές υποχρεώσεις, που είναι δεσμευτικές για τα κράτη-μέλη της Ένωσης. σε οποιοδήποτε πλαίσιο και αν εφαρμόζονται αυτές, του ΟΣΑ, του ΟΗΕ, της Ένωσης, είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι σημαντικό νομίζω να πούμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να προωθηθούν, πρέπει να ελέγχονται αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από τα του οίκου μας για να περάσουμε μετά σε διεθνές επίπεδο. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πολλές φορές δεν έχει υπάρξει η επαρκής ε, δικαιο... Ε, λογοδοσία. Και είναι δεσμευτικά όλα αυτά και για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ακόμη και για τις ιδιωτικές εταιρείες. Βέβαια, το ερώτημα αυτό που έθεσε και ο Ρίτσαρντ. Δεν θέλουμε να διαδίδονται, να πλαπλασιάζονται αενάως οι ύπατοι εκπρόσωποι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και χρήσιμο τελικά να υπάρχει ένας τέτοιος εκπρόσωπος. Οπότε σκεφτείτε το. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ποπόφσκι μπορεί να μας πει κάτι παραπάνω. Αν υπάρχει κάτι που να είναι στα σκαριά ως προς αυτό. Και τέλος, είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα πλαίσια να εξασφαλίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα λαμβάνονται πάντα υπόψη σε όλη τη διαδικασία λήψη απόφαση στο Συμβούλιο. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί αυτό μέχρι στιγμή. Νομίζω ότι έχει υπάρξει ένα τρομακτικό έλλειμμα. Υπάρχουν πολιτικές ε, κάποιων χωρών που έχουν ε, παραμελήσει εντελώς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε σας ρωτώ, η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων πιέζει για το PSE και για άλλους φορείς, οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα ανθρώπινα δικαιώματα στην χάραξη πολιτικής και βεβαίως στις περιπτώσεις ε, παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μας πει ο κύριος Ποπόφσκι την άποψή του. Ε, ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλες τις ε, Πληροφορίες που ο Υπουργός κ. Ποπόφσκι μας ε, παρουσίασε επίσης ε, ε, Χαίρομαι που παρά τις πολυάριθμες υποχρεώσεις σας προλάβατε να έρθετε να μας επισκεφθείτε. Θα ήθελα τώρα να αναφέρω δύο θέματα που προέκυψαν. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία. Είπατε ότι δεν είναι απόλυτα σαφές ε, κατά πόσο αυτό το μέσο θα ε, αποτελεί πραγματικότητα μέχρι τα τέλη του έτους. Ε, στη συνεδρίαση της υποεπιτροπής μας συχνά συζητούσαμε για αυτό το θέμα. Ορισμένοι από εμάς είχαν ερωτήσεις. Άλλοι αναρωτιόνταν κατά πόσο αυτό το μέσο θα παρέχει προστιθέμενη αξία. Εγώ ανήκω στην ομάδα που υποστηρίζει αυτή την πρωτοβουλία επειδή πιστεύω ότι η δραστηριότητα των υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διάφορες χώρες ε, δείχνει ότι η δική μας αντίδραση των ε, ευρωπαϊκών οργανών είναι πολύ αργή. Σήμερα, για παράδειγμα, στη Λευκορωσία έχουμε πολλά φορέους, πολλά ιδρύματα που λειτουργούν ικανοποιητικά και που χρειάζονται χρήματα και τα ταμεία μας ε, ενεργοποιούνται πολύ αργά και αυτοί χρειάζονται αυτά τα χρήματα αμέσω ώστε να επιβιώσουν. Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε ότι ορισμένε χώρες εξακολουθούν να έχουν αμφιβολίες όσον αφορά αυτή την πρωτοβουλία. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή Αυτές οι αμφιβολίες, αυτές οι παρατηρήσεις είναι ουσιώδους ε, σημασίας, ε, είναι επί της ουσίας ε, επί της ύπαρξης αυτού του μέσου ή πρόκειται για απλά τυπικές ερωτήσεις. Επειδή εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων. Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω πρόκειται για θέματα πολύ σημαντικά που ανέφεραν η κυρία Γκόμης και ο κύριος Χαουίτ για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που εξακολουθεί να εξελίσσεται Είπατε ότι οι υπευθύνοι αυτή τη υπηρεσία θα ε, μάθουν καλύτερα την ευρωπαϊκή δράση, αλλά εμεί θέλουμε να προχωρήσουμε πιο κάτω. Σε ορισμένες χώρες ε, στις πρεσβείες που υπάρχουν σε ορισμένε χώρες θα πρέπει να δημιουργηθούν μονάδες οι οποίες θα ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, ειδικευμένε μονάδες. Σε ορισμένες χώρες λοιπόν, σε ορισμένε χώρε θα πρέπει να προβλεφθούν αξιωματούχοι επαφή οι οποίοι θα διατηρούν την επαφή με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Θέλουμε να περιοριστούμε σε μόνο γενική εκπαίδευση, κατάρτιση ή πραγματικά θέλουμε να εκπαιδεύσουμε διπλωμάτες ε, οι οποίοι θα έχουν αυτό το ζήτημα ως ε, κύρια αποστολή. Ευχαριστώ. Presidente, eu creio Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι τρεις τελευταίοι ομιλητές κάλυψαν πολλά από τα πράγματα που θα ήθελα να αναφέρω. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ, τόσο όσον αφορά την ε, ευθυγράμμιση των δράσεων ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να ε, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι όλων των πολιτικών μας και όλων των ζητημάτων που εξετάζουμε. Για παράδειγμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να εντάσσονται στις, ε, συμφωνίες, στις εμπορικές μας συμφωνίες, στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης μας και ούτω καθεξής. Το ερώτημα είναι δεν θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό ε, πιο αυστηρά από ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα. Όσον αφορά τώρα τα δημοσιονομικά μέσα για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία, εδώ πιστεύω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο από ότι σήμερα. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία, ε, επικροτώ αυτή την ιδέα, όπως και ο κ. Χάουιτ, αλλά ε, αυτή η ιδέα δεν αρέσει σε όλα τα μέλη αυτού του κοινοβουλίου. Όπως είπε και ο κύριος Ζέμκε, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ε, αμφισβητούν, ε, έχουν ενδιασμού για τα οικονομικά θέματα αυτού του ευρωπαϊκού μέσου. Πιστεύω λοιπόν ότι μέλη αυτού του κοινοβουλίου όπως εγώ θα σας ήμασταν υποχρέοι αν μπορούσαμε να έχουμε μια ισχυρότερη γνώμη όσον αφορά αυτό τον οργανισμό. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά και να έχει και κάποιο βαθμό ελέγχου ε, στον τρόπο διαχείρισης αυτού του μέσου. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μια γενική εικόνα ε, του τρόπου δαπάνη των κονδυλίων που θα θεωρηθούν σε αυτό το μέσο. Ειδικότερα έχω ακούσει κάποιες ε, ενδιασμούς ε, όσον αφορά τις οικονομικές πτυχές από κάποια κράτη-μέλη. Επίσης τίθεται το ερώτημα των διπλών προτύπων, των διπλών στάνταρ. Ο τρόπος που χειριζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα διπλά στάνταρ, αυτό αποτελούν ένα φαινόμενο που υπαρκτό θα έλεγα. Μου φαίνεται ότι είμαστε πολύ άκαμπτοι όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου μας. αλλά δεν είμαστε τόσο αυστηροί όσον αφορά τις παραβιάσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατά ορισμένων προσφύγων. Για παράδειγμα, και αυτό φυσικά ε, δεν κάνει καλό στην εικόνα μας ε, σε όσους προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε με τις, ε, τα ψηφίσματά μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, η Επιτροπή Αναφορών και άλλα σώματα θα πρέπει να εξασκήσουμε κάποια πίεση ώστε να εξαλείψουμε αυτά τα διπλά στάνταρ. Επίσης έχω και μια συγκεκριμένη ερώτηση για εσάς. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με τα αρχικά εγγραφά που συντάξατε όσον αφορά το βαθμό στον οποίο η Υπηρεσία εξωτερική δράση θεωρεί ότι θα έπρεπε να συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για τις εξωτερικές υποθέσει. Η ανησυχία μου εδώ Η ανησυχία μου εδώ είναι ότι δεν θα έχουμε αρκετά ε, ισχυρή επιρροή σε θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί τι πράττει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρία Γκόμες, η ερωτήση μου προς ε, τον κύριο Ποπό. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία, εγώ είμαι ένα από τους ανθρώπους που το υποστηρίζουν. Ήμουν από τους πρώτους ε, που υποστήριξε αυτήν την άποψη το 2012 την ιδέα ότι θα δημιουργίας αυτού του μέσου διότι διαβλέπω καθαρά την ανάγκη να υποστηρίξουμε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να βοηθήσουμε στη δημιουργία οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία σε πολλά μέρη του κόσμου και όχι μόνο στην, στους ανατολικούς γείτονές μας όπως φαίνεται να είναι σήμερα το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογή ε, αυτού του μέσου. Συζητήσαμε τις προάλλες ε, στην Επιτροπή ΑΦΕΤ ε, όπου αναφέρθηκαν δύο πράγματα τα οποία με ανησυχούν στις κατευθυντήρες οδηγίες που πρόκειται να εγκριθούν όπως άκουσα από το Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα νομίζω ή σύντομα τέλος πάντων ειδικότερα η αξία αυτού του μέσου είναι ότι συνιστάται στο γεγονό ότι θα είναι ευέλικτο και ταχύ ότι θα διατίθενται άμεσα γρήγορα τα κονδύλια για αυτό το λόγο δεν μπορεί να έχει δομή διακυβέρνηση όπου κάθε κράτος μέλος ε, που συμβάλλει θα παρίσταται, δηλαδή 27 κράτη-μέλη, αυτό θα αποτελούσε υπερβολικό φόρτο. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να φροντίσουμε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα της Ευρώπης όπως ε, αντιπροσωπεύεται σε αυτό το κοινοβούλιο να αντιπροσωπεύεται και εκεί στο Συμβούλιο Διακυβέρνησης, στο Διοικητικό Συμβούλιο του μέσου αυτού. Και φυσικά καμία δράση δεν θα εγκρίνεται χωρίς συνένεση σε αυτό το πλαίσιο. Αντί λοιπόν έχουμε έναν αντιπρόσωπο από το Συμβούλιο, έναν από την Κομισιόν και έναν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και αντιπροσώπευση του Κοινοβουλίου που θα καλύπτει ολόκληρο ε, το εύρος. Αυτό θα ήταν μια καλή αντιπροσώπευση αντί για αντιπροσώπους που εκφράζουν τις απόψεις του κάθε κράτους μέλους. Ο τρόπος κινητοποίησης κονδυλίων εάν πρόκειται να πάρουμε χρήματα από οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα μέσα θα έπρεπε να είναι το μέσο δημοκρατίας και ανθρωπινών δικαιωμάτων διότι είναι ήδη υπαρκτό έχει ήδη το πεδίο δράσης του τα χρήματα δεν θα πρέπει να λυθούν από αυτό θα πρέπει να λυθεί από άλλα μέσα όπου υπάρχουν υπερβολικά πολλά χρήματα και όπου δεν λαμβάνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα υπόψη όπως ας πούμε το μέσο σταθερότητας Ελπίζω ότι θα μπορούσατε να το λάβετε υπόψη σας. Ευχαριστούμε. Δεν ε, βλέπω να έχει ζητήσει άλλο το λόγο εδώ, οπότε θα μιλήσω εγώ. Πρώτα απ' όλα, η στρατηγική αυτή έχει να κάνει με το 2010. Νομίζω ότι το γεγονός ότι τόσο αργά μιλάμε για την έκθεση αυτή του 2010 και ότι θα παραταθεί κι άλλο η διαδικασία δεν είναι κάτι θετικό. Ξεχνάμε τα γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα. Ξεχνάμε τα γεγονότα τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν στην εξέταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό και πρέπει να επιταχύνουμε τον ρυθμό εξέτασης. Δεύτερον, ο υπουργό το επιβεβαίωσε επίσης. Οι εργασίες για τη νέα στρατηγική όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα προκάλεσαν πολλές συζητήσεις και ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στην υποπιτροπή μας και την είπα το εκπρόσωπο. Ελπίζω το Δεκέμβριο στη συνάντησή μας να καταλήξουμε σε ένα προϊόν, σε ένα αποτέλεσμα το οποίο να αποτελέσει και συμβιβασμό ανάμεσα στην ΕΠΑ, το εκπρόσωπο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Δημοκρατία, το Ευρωπαϊκό αυτό μέσο, πιστεύω ότι όλοι κατανοούμε πως είναι κάτι αναγκαίο. Σήμερα το μέσο που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό. Για την περίπτωση της Κούβας, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τέτοιου είδους χώρες με αυτό το μέσο. Δεν είναι αποτελεσματικό. Χρειαζόμαστε άλλα μέσα πιο ελαστικά. μέσα τα οποία να μην συνοδεύονται από τεράστια γραφειοκρατία στη χώρα μου, λέμε συχνά ότι αυτός που δίνει γρήγορα δίνει το διπλό. Η διαδικασία αυτή καθεαυτή μπορεί να βλάψει τις πρωτοβουλίες οι οποίες γεννιόνται μέσα σε μια τέτοια χώρα. Είναι Κάτι που παίρνει μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα τώρα που βρισκόμαστε εν μέσω της Αραβικής Άνοιξης. Πρέπει συνεπώς να βρούμε τον καλύτερο τρόπο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να υπάρχει ένα τέτοιο μέσο πάντως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, να προσπαθήσω να απαντήσω στις ε, ερωτήσεις σας, λέει ο κύριος Ποπόφσκι για τόσα αναφέρονται στην επιστολή στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Χόουιτ. Ναι, τα αναγνωρίζουμε, τα λαμβάνουμε υπόψη και θα τα συμπεριλάβουμε όταν τελειώσουμε την πρόταση και είμαστε έτοιμοι για τη συζήτηση. Είναι αλήθεια ότι επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στη διαδικασία. Γιατί, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει τώρα να στραφούμε και στο περιεχόμενο. Και ελπίζω και πιστεύω ότι το περιεχόμενο τελικά και η συζήτηση θα αποτελούν ένα καλό σημείο κίνησης. Η διαδικασία θα συνεχιστεί. Δεν θα μείνουμε όμως στη διαδικασία. Χρησιμοποιούμε τη διαδικασία για να μιλήσουμε για το περιεχόμενο στο Συμβούλιο πρέπει τα κράτη-μέλη να πούν την άποψή τους. Να δούμε πώς σκοπεύουν να συνεισφέρουν έτσι στη πολιτική μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι πιο αποτελεσματική. Εσείς αναφερθήκατε βέβαια σε διάφορα ειδικά ζητήματα. Για τον ειδικό εκπρόσωπο. ή ο εκπρόσωπος δεν σκοπεύει να προτείνει έναν ειδικό εκπρόσωπο. Σημείωσα τα σχόλιά σας. Όπως ξέρετε, μέχρι τώρα ε, το USR είναι ένα μέσο εξωτερικής πολιτικής. Το Συμβούλιο έχει ειδικού εκπροσώπους για ορισμένες χώρες της περιοχής. Ποτέ δεν είχε ειδικού εκπροσώπους για ένα θέμα. Για χώρες, ναι. Μπορεί να είχαμε στο παρελθόν ειδικού που είχε ορίσει ο Χαβιέρ Σολάνα, αλλά και πάλι ήταν ένα διαφορετικό επίπεδο συμμετοχής μας. Ήπατος εκπρόσωπος λοιπόν δεν σκοπεύει να προτείνει κάτι τέτοιο. Ευχαρίστως όμως να το συζητήσουμε μαζί σας. Αυτά που είπατε για τη διεθνή δικαιοσύνη φυσικά και ισχύουν. Διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακριβώς αυτή είναι μια από τις αδυναμίες μας, η αποτελεσματικότητα. Θα ήταν κάπως παρακινδυνευμένο να υπάρχει διακοπή. Ακόμα και αν ο διάλογος πάει καλά, συγχρόνως εμείς πρέπει να ξέρετε ότι ολοκληρώνουμε το σχετικό διάλογο με τη Ρωσία. Συνήθως το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό. Θα ήταν όμως φάλμα να πούμε πως όχι, δεν θα το κάνουμε πια. Πρέπει να σκεφτόμαστε δυο φορές πριν αποφασίσουμε για να δούμε πώς, με ποιο τρόπο θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Πάντως όταν ερχόμαστε στην εσωτερική οργάνωση, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ξεκινάμε επιστήνοντας την προσοχή των συναδέρφων από διάφορες υπηρεσίες. Να πούμε ότι δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην γεωγραφική ε, μορφή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε την Τρίτη Επιτροπή για παράδειγμα για την Κίνα. Εκεί έγινε μια σημαντική συζήτηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε ενία θέση. Δεν συμβαίνει όμως πάντα. Τα μέσα στα οποία αναφέρεστε λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Μέσο για Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα θα συνεχίσει, θα αποτελεί πακέτο των δημοσιονομικών μέσων για το, την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Θα συζητηθεί και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στις αρχές της επόμενης χρονιάς νομίζω. Και η διαδικασία θα είναι σημαντική, γιατί το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ξεκινούν να συζητούν τα μέσα και συγχρόνως στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην Κομισιόν θα ξεκινήσει η προετοιμασία του νέου δημοσιονομικού κύκλου. Είναι και αυτή μια ευκαιρία για να λάβουμε περισσότερο υπόψη μας οριζόντια ζητήματα όπω είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να σκεφτούμε δηλαδή λίγο πιο πέρα από του στόχου του Ευρωπαϊκού Μέσου για Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, γιατί μπορεί να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέσα. Να βρούμε δηλαδή άλλες δράσεις, DCI, DF κλπ. Μόλι ξεκινήσαμε τη δουλειά και για κατευθυντήριε γραμμέ. Ε, προγράμματος, κάτι το οποίο ετοιμάζουμε με την Κομισιόν. Είναι μια μοναδική ευκαιρία αυτή να σκεφτούμε τέτοια οριζόντια ζητήματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα από αυτά. Ένα άλλο είναι η σχέση ασφάλειας και ανάπτυξης. Είναι ένα διαφορετικό θέμα αυτό βέβαια. Θα επανέλθω αργότερα στο μέσο για τη δημοκρατία. Προσπαθώ να είμαι σύντομος. Η ύπατος εκπρόσωπος φυσικά και θέλει να δώσει τη δικιά της άποψη και έρχομαι τώρα στην κυρία Γκόμες το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια όπως σας είπα. Η διαδικασία και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο έχει μεγάλη σημασία. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι ένα μέσο. Γι' αυτό και μας πήρε πολύ καιρό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επίτροπο Μάλστρομ, την Επίτροπο Ρέντινγκ και τους υπόλοιπους που έχουν λόγο γι' αυτά. Είναι, είναι θέμα ε, αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το παίρνουμε πολύ στα σοβαρά αυτό. Τώρα, ο ρόλος των κρατών μελών. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται πάρα πολύ να δώσουν συνέχεια στην πρόταση και ορισμένοι είναι πραγματικά πρωταθλητές στα ανθρώπινα δικαιώματα και μας πιέζουν να προχωρήσουμε με τις προτάσεις μας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πιέσουμε το Συμβούλιο. Ε, το θέλει. Αλλά όπως είπα, οι συζητήσεις άργησαν να ξεκινήσουν και κράτησαν πολύ για καλούς λόγους. Ήταν όμως ιδιαίτερα εντονές. αναφέρθηκα στη συζήτηση που θα έχουμε για τα οικονομικά μέσα. Για την ερώτηση του κυρίου Τάβαρη τώρα για τα οικονομικά μέσα και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα γίνει αυτό. Θα ισχύσουν οι κανόνες της Λισαβόνας. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, αλλά πολύ σημαντικές. Και ελπίζω ότι θα ξεκινήσουμε γρήγορα. Οι διαπραγματεύσει βέβαια θα πάρουν μέχρι τα μέσα του 2012. Η συζήτηση όμω για τα οικονομικά μέσα πρέπει να ξεκινήσει τώρα. Έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία, European Endowment. Δεν νομίζω ότι καμία χώρα είναι κατά Μπορεί να έχουν πράγματα να ρωτήσουν, να βάζουν κάποια θέματα, αλλά δεν αντιτίθεται στην ιδέα. Και συμφωνώ με αυτό που λέτε κι εσείς, ότι χρειαζόμαστε ένα σώμα, δεν είναι ένα θεσμικό όργανο, χρειαζόμαστε όμως κάτι το οποίο να είναι πιο ελαστικό και να μπορεί να κάνει ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε με τα ήδη υπάρχοντα μέσα. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Εγώ δεν είμαι ειδικό σε δημοσιονομική ε, management, αλλά να ξέρετε ότι όταν μιλήσαμε για τη γεωγραφική διάσταση, ήρθαν πολλές παρατηρήσεις που λέγανε ποια είναι τα λάθη που κάνουμε, δηλαδή ποιες χώρες μπορούμε να φτάσουμε. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, χρήματα ε, που είναι για άλλο σκοπό, για οργανώσεις που δεν είναι κατακαιγραμμένες, για παράδειγμα. Το θέμα της γεωγραφικής κάλυψης ήταν ένα ζήτημα. Και ο Πολωνός υπουργό και η κυρία Άστον έστειλαν ε, επιστολή πάντως στους υπόλοιπους υπουργούς ενημερώνοντας για την πρωτοβουλία και θυμίζοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσει. Συνεπώς, η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Είναι εφικτό αυτό. Κάποιο είδους γενική συμφωνία στο Συμβούλιο, δεν ξέρω. Είμαι όμως σίγουρος ότι το πρόγραμμα θα, έχει, θα μπορεί να ξεκινήσει τα μέσα της χρονιάς. γιατί η γεωγραφική κάλυψη δεν είναι για την ανατολική γυτνίαση. Ξεκίνησε από τη συζήτηση για την πολιτική γυτνίαση, αλλά ισχύει και μάλλον και στην αρχή ίσχυε μόνο για ανατολικά και νότια. Και μετά μπήκε το θέμα της χρηματοδότησης και συζητήσαμε σε βάθος με την Κομισιόν δεν πρόκειται τίποτα να αφαιρέσουμε από το IHR. Υπάρχει κάποιο περιθώριο στο μέσο γειτονίασης που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για δράση στην περιοχή, σεβόμενη τη γεωγραφική ισορροπία. Και αν λειτουργήσει και αν αποδειχτεί ότι αξίζει, μπορεί και να επεκταθεί περισσότερο. Θα μπορούσαμε δηλαδή να ψάξουμε να βρούμε άλλες πηγές από άλλα υπάρχοντα μέσα. Όχι όμως τώρα, ας ξεκινήσουμε πρώτα έτσι. Ας δούμε ποιες είναι οι ανάγκες που πιέζουν περισσότερο στην περιοχή και μετά πάμε πιο πέρα και στο νότιο τμήμα. Δεν αποκλείουμε τίποτα. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φυσικά και είναι πολύ σημαντικός. Και κάτι σημαντικό για την κυρία που το είπε και στους υπουργούς είναι το εξή. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγάλη γραφειοκρατία. Θέλουμε να έχουμε ένα διοικητικό σώμα όπου θα συμμετέχουν κράτη-μέλη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπατος εκπρόσωπος και κοινοβούλιο. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Πρέπει να συζητήσουμε ακριβώ με ποιο τρόπο θα γίνει, αλλά εννοείται ότι πρέπει να εκπροσωπείται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αν έχουμε κάτι πιο μεγάλο, δεν ξέρω, εδώ δεν θα είναι εκτελεστικό αυτό το σώμα. Θέλουμε μια μικρή εκτελεστική επιτροπή, η οποία να διαχειρίζεται τα προγράμματα. Αλλά κάποιο πρέπει να έχει και την πολιτική εποπτεία και να ασκεί και τον δημοσιονομικό έλεγχο κυρίως για τα κονδύλια που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι βάζουν τα κράτη-μέλη, αυτά θα πρέπει να υπακούν στους εθνικούς κανόνες. Πάντως, θα φροντίσουμε να υπάρχει διαφάνεια σε ό,τι κάνουμε. Και θα λογοδοτούμε απέναντι στους φορολογούμενους. Για τον τρόπο λειτουργίας νομίζω ότι είπα ήδη η ταχύτητα, η ελαστικότητα είναι πράγματα τα οποία μας νοιάζουν. Θέλουμε να είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται Αλλιώς δεν έχει νόημα να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μέσο. Και οποιαδήποτε επικάλυψη βέβαια είναι προς αποφυγή. Να απαντήσω λίγο και σε αυτό που ρώτησε ο πρόεδρος για την ετήσια έκθεση. Ναι, σίγουρα πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα. Καθυστερήσαμε όχι μόνο εξαιτίας της δημιουργίας της ε, υπηρεσίας, αλλά μετέχαμε και την Αραβική Άνοιξη. Καθυστερήσαμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο μέλλον για να αποφεύγουμε τέτοιου είδου καθυστερήσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Ποβόφσκι. και για την εισαγωγική σας παρέμβαση και για τις απαντήσεις που δώσατε σε σχέση με τη στρατηγική σε σχέση με το μέσο για τη δημοκρατία. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και άλλες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Έχουμε καθυστερήσει λιγάκι, βέβαια. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Αίγυπτος. Ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με, την, με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου και τις εκλογές στην Αίγυπτο. Η Επιτροπή μας συχνά κάνει ανταλλαγές, πληροφο... ε, πληροφοριών και απόψεων με ε, εκπροσώπους σχετικά με την Αραβική Άνοιξη. Θα υπάρξει και συγκεκριμένη θέση από την Επιτροπή μας. Ε, σήμερα θα συνεργαστούμε με την ε, αντιπροσωπεία για το ΜΑΣΡΕΚ και παρακαλώ καθίστε. Η κυρία Μαρίζα Ματίας είναι μαζί μας. Nie wyrażał Parlament swoje obawy. E, są e, rezolucje. Βεβαίως μιλούμε και για την ε, καταπίεση μετά την ε, πτώση του Μουμπάρακ. Ε, έχει υπάρξει περιορισμός των ελευθεριών, η το ότι έχουν πάει πολλοί πολίτες ενώπιον δικαστηρίων είναι επίσης ένα θέμα που πρέπει να μελετήσουμε. Από τις 17 Νοέμβρη έχουν γίνει πολλές ε, έτσι, έχουν υπάρξει πολλές ε, διαμάχες μεταξύ των ε, δυνάμεων ασφαλείας, των διαδηλωτών. Στο Κάιρο, σε σχέση και με τις εκλογές, ο Μοχάμετ Ελμπαραντέι, ο πρώην πρόεδρος της ε, Διεθνούς Επιτροπής για την ε, Πυρηνική Ασφάλεια, έχει παρέμβει. Έχουν υπάρξει ε, χτυπήματα των δυνάμεων ασφαλείας που έχουν οδηγήσει σε θανάτους, σε τραυματίες. Πολλοί, έχουν, πολλοί δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί, έχουν βασανιστεί. Έχουν υπάρξει λοιπόν πολλές παραβιάσεις δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρουμε ότι κάποιοι θέλουν να παραταθούν, να αναβληθούν προς το παρόν οι εκλογές. Ο πρώτος γύρος έγινε χτες στις 28 ε, Νοέμβρη. Είναι σημαντικό λοιπόν να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία. Έχουμε και τον εκπρόσωπο του, την εκπρόσωπο της, ε, του δικτύου Euronet. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σα ενημερώσω πρώτα απ' όλα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο σήμερα. Πρέπει να περάσουμε στο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών συστάσεων από μέρου μα σήμερα. Η κατάσταση στην Αίγυπτο είναι κρίσιμη. Αντιμετωπίζουμε σημαντικά διακυβεύματα μετά από την επανάσταση της 25ης Ιανουαρίου του 2011 όπου οι άνθρωποι ζήτησαν το σεβασμό της ελευθερίας, της ε, ελευθερίας τους ε, σήμερα έχουν ξανακατέβει οι ίδιοι άνθρωποι στο δρόμο και διαδηλώνουν ώστε να ε, ε μην απογοητευτούν οι ελπίδες τους μην... Ε, υπάρχουν, έχουμε ακούσει καταδίκες για μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων από το Συμβούλιο των Στρατιωτικών Δυνάμεων γίνονται πιο συστηματικά ακόμη και από, από ό,τι συνέβαινε υπό το καθεστώς του Μομπάρακ έχει διευρυνθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πάνω από 12.000 δίκες έχουν λαβεί χώρα στα στρατιωτικό δικαστήρια. Ε, χρησιμοποιούνται συχνά, χρησιμοποιείται συχνά βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών και επιθέσεις κατά ε, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω ε, εκστρατιών ε, δυσφήμισης ε, ε, των μη και δημοσιογράφων, δικαστικές αγωγές κατά οργανισμών που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Διαπιστώνουμε επίσης περιθωριοποίηση του ρόλου των γυναικών στην πολιτική διαδικασία και πολλές παραβιάσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών. Σήμερα πολλοί ακτιβιστές και blogger έχουν μπει στη φυλακή όπως ο Μικελ Ναϊμπίμ καμία ανεξάρτητη έρευνα δεν προβλέπεται σήμερα όσον αφορά τα γεγονότα στα οποία αναφερθήκατε για τα γεγονότα που συνέβησαν στη διαδήλωση των κοπτών στο Κάιρο Υπάρχει μια εκθέση που τεκμηριώνεται από τους ε, ΜΚΟ και ήθελα να αναφερθώ σε ένα έγγραφο που προσπογράφεται από 12 οργανισμούς ε, της 25 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, το Ανώτατο Συμβούλιο των Στρατιωτικών Δυνάμεων αρνείται να συμμετέχει και έχει αποκλείσει τις ε, ομάδες νέων και, τις, ε, και τους οργανισμούς υπέρασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ και 10 μέρες. Οι διαδηλωτές που επιθυμούν περισσότερη δημοκρατία από οποιοδήποτε ε, τάξη της κοινωνίας διαδηλώνουν όχι μόνο στην πλατεία Ταχρήρα αλλά και στις υπόλοιπες ε, πόλεις της χώρας. Ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν αυτές οι ε, το νέο κύμα διαδηλώσεων που ξεκίνησε την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου είναι ένα έγγραφο το οποίο ψηφίστηκε για να ε, εξασφαλίσει συνταγματικά ε, δικαιώματα ε, περισσότερα από τα συνταγματικά στην εξουσία. Ζητούν λοιπόν να παραδώσει την εξουσία, η στρατιωτική εξουσία σε μια κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα ήταν χρήση βίας κατά των ειρηνικών διαδηλωτών. Σήμερα αντιλαμβανόμαστε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις διαδηλώσεις στην Αίγυπτο. Οι δυνάμεις ασφαλείας και οι στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και ε, πραγματικά πειρά. Πολλοί διαδηλωτές και πολλοί ε, δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί 41 πάνω από 3.000 τραυματίες ηλικίας μεταξύ 15 και 30 ετών και τύφλωση πολλών ατόμων ε, όλα αυτά έχουν καταδικαστεί από πολλούς ΜΚΟ από τα Ηνωμένα Έθνη Έχουμε λοιπόν εδώ κατάφορες ε, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι ΜΚΟ φοβούνται ότι το σημερινό κλίμα θα παρεμποδίσει το έργο τους ε, ε καταγγελίας των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ε, αδυναμία δημοκρατικών ε, εκλογών στην Αίγυπτο. Ως Ευρωπαϊκή, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, λυπούμαστε που δεν συμμετείχε ε, ως παρατηρητής στις εκλογές, όπως έγινε στην Τινησία. Υποστηρίζουμε επίσης ορισμένα σημεία τα οποία ανέφερε η υπατή εκπρόσωπος της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την... όπως την ελευθέρωση των διαδηλωτών, το, ε, την παράδοση της εξουσίας σε μια ε, κυβέρνηση αιρετή. Η υποβάθμιση αυτή της κατάστασης των ανθρωπινών δικαιωμάτων ε, δεν έλαβε την κατάλληλη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα ένα σαφές και δυνατό μήνυμα κατά των παραβιώσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρούμε ότι σήμερα πρέπει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασκήσει πίεση ισχύρη ώστε να αποφευθεί η κλιμάκωση της, ε, στρατι... της καταπίεσης και ε, ώστε να περάσουμε σε μια αιρετή κυβέρνηση. Εν ώψη του επόμενου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα λάβει χώρα την 1η Δεκεμβρίου θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στις αρχές της μεταβατικής αρχής της Αιγύπτου την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ζητήσουμε την άμεση διακοπή της χρήσης ε, μέσων βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, την διεξαγωγή αμερόληπτων ερευνών κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά από την πτώση του καθεστώτος του Μουμπάρακ, την τήρηση της ελευθερίας έκφρασης του συνεταιρίζεστε και της ε, ειρηνικής διαδήλωσης και του τύπου. Επίσης να σταματήσουν οι διαδικασίες δυσφήμισης για τους καπαόψιλων στις ε, κρατικές εκστρατείες. Σήμερα υπάρχει πραγματικός κίνδυνος όσον αφορά τη μελλοντική δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδότηση των οργανισμών υπερέψης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Επίσης θέλαμε την απελευθέρωση όσων φυλακίστηκαν για την απλή συμμετοχή τους σε, διαδηλώσεις, σε ειρηνικές διαδηλώσεις. Όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ζητήσει από τις Αιγυπτιακές Αρχές να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών για τις, ε, όπως ονομάζουμε, μεταβατικές αποφάσεις. Τέλος, η ευρωπαϊκή πολιτική υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορέσει να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο μόνο αν συνοδεύεται από πολιτική υποστήριξη και όχι μόνο οικονομική. Δεν μπορούμε να παραμένουμε θέατες των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στην Αίγυπτο. Χρειάζεται πολιτική υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των δημοκρατικών δυνάμεων στην Αίγυπτο. Αυτή είναι η νέα προσέγγιση που θα πρέπει να έχουμε στο πλαίσιο της νέας πολιτικής γειτονίας για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έχει μια ιστορική ευκαιρία να αποδείξει την πολιτική της βούληση και την αξιοπιστία της υλοποιώντας μια νέα πολιτική αποτελεσματικής και πραγματικής υποστήριξης της δημοκρατίας σε όλες τις χώρες του αραβικού κόσμου. Για να ολοκληρώσω. πολλές φορές έχουν διατυπωθεί ε, συστάσεις για την Αίγυπτο και για τις υπόλοιπες χώρες. Πιστεύουμε ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντικός ε, για την υπερασπίση των ε, ΜΚΟ. Επίσης καλούμε τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μεταβούν στην Αίγυπτο να συναντήσουν την κοινωνία των πολιτών και να αντιληφθούν την κατάσταση στην ίδια τη χώρα. E, Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Μαρίζα Ματίας, την πρόεδρο της αντιπροσωπείας για τις χώρες του Μασρέκ. Ευχαριστώ. Πολλά από όσα ήθελα να πω υπόθηκαν ήδη. Οπότε ίσως ε, έτσι κάποια δεδομένα θα ήθελα απλώ να σας ε, αναφέρω ε, για πράγματα που συνέβησαν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στο Κάιρο για το ποια είναι η κατάσταση δηλαδή που επικρατεί πλέον στην Αίγυπτο. Υπάρχει μεγάλη ένταση, υπάρχει ένα είναι σαφές έτσι το ότι υπάρχει ένταση μεταξύ των δημοκρατικών δυνάμεων που έχουν την εξουσία και που θέλουν να παραμείνουν στην εξουσία και όσων ε, είναι αντίθετοι. Ήμουν εγώ στο Κάιρο, όπως σας είπα. Ε, δεν μπορούσαμε βεβαίω να πλησιάσουμε όλες αυτές τις, όλα αυτά τα σημεία στην πόλη. Ε, μπόρεσα όμως να μιλήσω με πολλούς εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, με εκπροσώπους της ε, αντιπολίτευσης. Και ήταν πραγματικά πολύ ιδιαίτερη η κατάσταση. Έχουμε λάβει ήδη θέση για το τι έχει γίνει. Έχουμε ψηφίσει ψηφίσματα. Και αυτό που, έχει, αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα είναι πραγματικά μια έκτακτη κατάσταση. Βρισκόμαστε τώρα σε μια διαδικασία εκλογική και ανεξάρτητα από το τι πιστεύουμε ιδεολογικά ή πολιτικά πρέπει όλοι νομίζω να πούμε ότι Έχει υπάρξει μια, ένα είδος έτσι, πνευματικής δικτατορίας στην ε, Αίγυπτο σε αυτές τις εκλογές. Ε, δεν είχα α, το, την δυνατότητα να είμαι εκεί στο κέντρο των εξελίξεων, αλλά είδα πώς οι άνθρωποι κινητοποιούνται και πώς δραστηριοποιούνται για όλη αυτή τη διαδικασία των εκλογών δεν το λέω βεβαίω τώρα εδώ για το είναι την προσωπία του Μασρέκ, αλλά είναι, αυτό που σας λέω είναι δική μου προσωπική άποψη. Ε, προφανώς δεν θέλουμε να εμπλακούμε αλλά, ή να παρέμβουμε, αλλά προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε και έτσι να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά για, τις, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του πληθυσμού ε, και πρέπει αυτή η δημοκρατική διαδικασία να γίνει χωρίς ε, προσκόμματα να διεξαχθεί χωρίς προσκόμματα. Βεβαίως, τις συνέπειες τις ξέρετε. Οι αρχές και το καθεστώς έχουν ε, προγραμματίσει ας πούμε την δυνατότητα το κοινοβούλιο να μπορεί να ελέγχει τις δαπάνες του προπολογισμού Προς το παρόν όμως έχουμε μια μεταβατική κυβέρνηση και αυτό που ε, βλέπουμε στην Αίγυπτο είναι ουσιαστικά ότι κυριαρχεί το Στατιωτικό Συμβούλιο, το οποίο εμένει σε κάποια προνόμια που είχε και θέλει να εξακολουθήσει να τα έχει. Διάφορα κόμματα, διάφορα μη κυβερνητικές οργανώσεις ζήτησαν οι εκλογές να προετοιμαστούν καλύτερα, έτσι ώστε να μην ξαναζήσουμε αυτό που έγινε στην Ινδονησία και αλλού. Είναι όμως πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό και αυτή η μεταβατική διαδικασία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το είδαμε τις τελευταίες ημέρες και στην ε, περίπτωση της δικής μας, τη δική μας, την, ε, της αντιπροσωπείας δηλαδή του Μασρέκ, δεν είχε ζητηθεί να γίνει η παρατήρηση εκλογών, δεν ήταν και δυνατόν ε, και δεν ήταν και η πρόθεσή μας. Η πρόθεσή μας ήταν να δείξουμε στην Αίγυπτο ότι χρειάζεται ένα δημοκρατικός εκλεγμένο κοινοβούλιο. Ένα αντίβαρο στην, ε, στο Στρατιωτικό Συμβούλιο. Βεβαίω είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά. Αυτή βεβαίως είναι δική μου άποψη προσωπική. Και βεβαίως δεν το θέμα δεν είναι να πάρουμε το μέρος του ενό ή του άλλου. Έχουμε μια εξαιρετική ε, κατάσταση, έκτακτη κατάσταση και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε και σαφή μηνύματα. Υπάρχει επιθυμία να υπάρξει δημοκρατία στην Αίγυπτο και αυτό θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Θα δούμε λοιπόν ε, προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι εξελίξεις. Όλα τα, πραγμα... όλα τα μέτωπα ακόμα είναι ε, ανοιχτά. Δεν ξέρουμε λοιπόν πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν διάφορα πολιτικά κόμματα, υπάρχουν πολλοί που θέλουν να είναι υποψήφοι, αλλά τελικά δεν μπόρεσαν. και υπάρχουν και πολλοί που, ε, έχουν, που είχαν θεμητά ε, συμφέροντα για να συμμετάσχουν, αλλά τελικά τους μπλόκαραν. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Γκόμε έχει ζητήσει το λόγο. να σας ζητήσω να είσαστε σχετικά σύντομοι. Ευχαριστώ. Άκουσα τι διπόθηκε και εκφράζω την πλήρη μου αλληλεγγύη προς όλους αυτούς που μάχονται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Αίγυπτο και που είναι αντιμέτωποι με ένα τέτοιο καθεστώς σκληρό. με τον τρόπο που δρά απέναντι στον πληθυσμό. Πιστεύω πως είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο μας να τοποθετηθούμε λέγοντας ότι οι εκλογές αυτές στην Αίγυπτο δεν μπορούν να θεωρηθούν εκλογές οι οποίες τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές. Διότι, εντάξει, εγώ πήγα 19 Μαρτίου που ήταν το δημοψήφισμα, δεν έχει καμιά σχέση, και είδα ότι ο πληθυσμός φυσικά και ήθελε να εκφραστεί, ήθελε να κάνει τη φωνή του να ακουστεί, ήθελε να φτιάξει μια σύγχρονη Αίγυπτο. Η αλήθεια είναι όμως πως η διαδικασία αυτή δεν οδήγησε για παράδειγμα σε παρατηρητές. Θα μπορούσαν να υπήρχαν πολύ περισσότεροι που να παρακολουθήσουν τις εκλογικές διαδικασίες στην Αίγυπτο. Άρα κάποιος πρέπει να βρει το θάρρος και να πει ότι παρόλα αυτά, παρά το τεράστιο ενδιαφέρον που δείχνουν οι Αιγύπτιοι για τη δημοκρατία στη χώρα τους, παρόλα αυτά θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το ποσοστό παρουσίας τελικά στις εκλογές αυτές. Οι εκλογές αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ε, πηγή νομιμότητας ενός κοινοβουλίου. Θα υπάρξει μια κοινοβουλευτική δομή βέβαια, προσωρινή, που θα οδηγήσει ίσως σε κάποια κυβέρνηση, μέχρι όμως να υπάρξουν πραγματικές εκλογές που να ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές. Ευχαριστούμε, ο κύριος ε, Κάζακ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να εκφραστώ εδώ και να μιλήσω για αυτού που παρεβαίνουν υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Δυστυχώ, μετά την πτώση του καθεστώτος του τέος Αιγύπτιου Πρόεδρου, Μουμπάρακ, ο Αιγυπτιακός λαός αξίζει περισσότερα. Μετά από τόσα θύματα οι Αιγύπτιοι αξίζουν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων των δημοκρατικών δυνάμεων, καθώς επίσης και την στήριξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όμως η μετάβαση αυτή έρχεται αντιμέτωπη με διάφορες δυσκολίες. Διαπιστώνουμε απουσία δημοκρατικών συνηθιών. Διαπιστώνουμε μάλλον χάος και δυσκολίες να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός μετάβασης προς τη δημοκρατία. Όμως παρόλα αυτά πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να βοηθήσουμε κι εμείς, ώστε να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών, τα μέσα ενημέρωσης, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, μια που διαπιστώνουμε πράξεις βίας σε βάρος των δημοσιογράφων, σε βάρος των μέσων ενημέρωσης. Όλα αυτά δεν δείχνουν βέβαια καλή θέληση από πλευράς των αρχών δεν δείχνουν ότι οι αρχές θέλουν πράγματι να πάνε προς τη δημοκρατία. Γι' αυτό και λέω ότι εμείς πρέπει να πιέσουμε δημοκρατικά, ευγενικά, αλλά να ασκήσουμε παρόλα αυτά πίεση απέναντι στις αρχές, ώστε οι Αιγύπτιοι της πλατείας Ταχύρ, να, της πλατείας Ελευθερίας, να καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους. Πρέπει να βοηθήσουμε τα κινήματα αυτά και οικονομικά Μάλιστα, είχαμε και μία πρόταση για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Θέλω να ευχαριστήσω πάντως όλους όσοι δουλεύουν υπέρ της αλλαγής και σας ζητάω να συνεχίσετε προς την ίδια κατεύθυνση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τώρα θέλω να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, τον κ. Ζάνα, να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Oui, après-midi. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε με όσα υπόθηκαν όσον αφορά την τραγωδία που συνέβη στους διαδηλωτές στην πλατεία Ταχρήρ αυτό το περιστατικό εξαιρετικής βίας στις 19 και 20 Ιανουαρίου όπου τόσα άτομα τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν. Το ζήτημα ε, σήμερα είναι ποιε ήταν οι εξελίξει μετά από τα ψηφίσματα που, που ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την Αίγυπτο. Δυστυχώ ε, σε πολλά μέτωπα διαπιστώνουμε ότι οι blogger παραμένουν στη φυλακή ότι η δυσανάλογη χρήση βίας και καταπίεση συνεχίζει παρότι αναγνωρίζουμε ότι τις τελευταίες μέρες οι στρατιωτικές δυνάμεις ε, ε, ε, επενέβησαν μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών της πλατείας Ταχρήρ για να σταματήσει η εξάσκηση βίας ε, προς τους διαδηλωτές. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν τραυματισμένοι, νεκροί και συλληφθέντες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες εξελίξεις θετικές μετά από αυτές τις διαδηλώσεις ε, για παράδειγμα μια υπόσχεση που παραμένει ωστόσο υπόσχεση απομένει να δούμε κατά πόσο θα την τηρήσουν οι στρατιωτικές αρχές για τη διεξαγωγή εκλογών πριν από τον Ιούνιο του 2012 επίσης η υπόσχεση ότι οι τρέχουσες έρευνες όσον αφορά τα γεγονότα και οι έρευνες για τον καθορισμό, για την αποδόση ευθυνών όσον αφορά τα γεγονότα του Νεμβρίου στην πλατεία Ταχρήρ Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η εξέλιξη είναι ευπρόσδεκτη από μέρους μας όσον αφορά τις πιέσεις που εξασκούμε καθημερινά ζητώντας ε, την άρση του νόμου ε, κατάστασης έκτασης ανάγκης η ε, υπατή εκπρόσωπος επίσης στην τελευταία της δήλωση της, του Νοεμβρίου υπογράμμισε και ζήτησε από τους στρατιωτικούς να έρουν το ταχύτερο δυνατό ε, το νόμο έκτακτης ανάγκης να επιτρέψουν τη, σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτά θα μεταφραστούν σε πραγματικά γεγονότα, θα υλοποιηθούν πραγματικά. Μια άλλη θετική εξέλιξη είναι η έναρξη των εκλογών που ξεκίνησε στις 28 Νοεμβρίου. Η πρώτη αναφορά που έχουμε λάβει από την αντιπροσωπεία, γιατί παρότι δεν τις παρατηρούμε επίσημα, έχουμε 50 διπλωμάτες εκεί συντονισμένους από τους διπλωμάτες του Καΐρου και έχουν πρόσβαση ε, και μας ανακοινώνουν ε, θετικά νέα. Υπάρχει λοιπόν ε, μια αισιοδοξία. Όσα έγιναν είναι καταδικαστέα, είναι τραγικά. Εξακολουθούμε τις πιέσεις προς τις Αιγυπτιακές αρχές ώστε να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και αυτό είχε θετικά αποτελέσματα διότι βλέπουμε ότι ε, σημειώνονται ουσιαστικές ε, εξελίξεις. Δίνω το λόγο στον συναδελφό μου του τμήματο που ασχολείται με την ε, παρακολούθηση των εκλογών. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις εκλογές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Μια σύντομη ενημέρωση σε σχέση με τις εκλογές από την αψή της παρακολούθησης. Όπως αναφέρθηκε σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι παρατηρητή των εκλογών. Ο λόγος είναι ότι δεν προσκληθήκαμε. Το ζήτημα πρόσκλησης του Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάστηκε πολλές φορές σε πολλά επίπεδα από την είπατε εκπρόσωπε, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το αναφέραμε το ζήτημα και σε διπλωματικό επίπεδο εδώ, ωστόσο οι Αιγυπτικές αρχές αποφάσισαν να μην καλέσουν κανέναν κρατικό οργανισμό όπως είπε ο συναδελφός μου, ε, συντονίζουμε ωστόσο τη διπλωματική παρακολούθηση στον τομέα αυτό και λαμβάνουμε εκθέσεις. Επίσης έχουμε ανοιχτό διάλογο με διεθνείς οργανισμούς που παρακολουθούν τις εκλογές. Επτά διεθνείς μη κυβερνητικοί οργανισμοί έχουν διαπιστευθεί επίσημα από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν διαπιστευτεί επίσημα, αλλά που τους έχει επιτραπεί η παρακολούθηση, όπως το NDI και το IRI της Αμερικής. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί είναι παρατηρητές και λαμβάνουμε αναφορές και παραμένουμε σε επαφή, όπως είπε ο συναδελφός μας, από την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μία αρκετά εμπεριστατωμένη άποψη του τι συμβαίνει, ότι η διαδικασία εξελίσσεται πολύ καλύτερα από ό,τι αναμενόταν από όλους και φυσικά συνεργαζόμαστε με τοπικούς παρατηρητές και έχουμε παρέχει χρηματοδότηση για την εκπαίδευση αυτών των παρατηρητών. Έχουμε δύο οργανισμούς με ε, ευρωπαϊκή ε, χρηματοδότηση που παρέχουν εκλογική υποστήριξη σε μικρόν για την υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι Πολλές φορές θα ξανασυζητήσουμε την κατάσταση στην Αίγυπτο. Σήμερα συζητήσαμε για αυτή τη δύσκολη διαδικασία που μόλις ξεκινάει και μιλήσαμε για την ε, καταστολή των διαδηλωτών από τις αρχές Ζητήσαμε και για το αίτημα αναστολή των εκλογών. Εξηγήσαμε ότι υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι στο πολιτική σκηνή. Δεν ζητούν όλοι την ε, αναστολή των εκλογών. Θα πρέπει πιστεύω να παραμείνουμε αισιόδοξοι. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι αλλαγές θα είναι μεγάλες και ότι το καθεστώς ε, στην Αίγυπτο θα αλλάξει. Ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους μας τους προσκεκλημένους, την κυρία Ματιάς κυρίως. Και θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο, καθώς έχουμε κάποια καθυστέρηση. Εδώ θα μιλήσουμε για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Σουαζιλάνδη. Ειδικότερα θα μιλήσουμε για τα δικαιώματα των γυναικών. Εδώ θα λάβουμε υπόψη την ε, καθολική περιοδική εξέταση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Πρόεδρος σε το μικροφόνο. Όσον αφορά την υποεπιτροπή μας, εφόσον συζητάμε για αυτό το ζήτημα, παρότι δεν πρόκειται για τόσο ε, σημαντική επικαιρότητα όσο η Αίγυπτος ή η Αραβική Άνοιξη. Η Σουαζιλάνδη δεν νομίζω ότι αποτελεί αντικείμενο οποιοδήποτε ψηφίσματο του Κοινοβουλίου, παρότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ ενισχυτική σε αυτή τη χώρα. Τουλάχιστον έτσι αυτή την εντύπωση σχηματίζουμε διαβάζοντα την έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το άτομο που ήθελα να καλέσω δεν είναι παρόν. Just Να συνεχίσουμε. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία πρόσωπο της, αμνηστι... της Διεθνούς Αμνηστίας και που έχει προετοιμάσει μια από τις εκθέσεις για τη Σουαζιλάνδη παρουσίασε αυτή την έκθεση στον υποτεκπρόσωπο των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Σας καλωσορίζω. English number two. Is okay? Mm-hmm. Yeah, but can you explain this? The first? Oh, you have to Introduce them. Oh, Przepraszam bardzo, mamy informację, że już mamy połączenie. Będziemy się łączyć. Θα ήθελα καλωσορίσουμε και τους προσκεκλημένους μας. Έχουμε μια βίντεο σύνδεση με την ε, Σουαζιλανδή. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Hans Willis Γέλε, και ο οποίο είναι πρόεδρος τη της ε, Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την κυρία Λαμίνη που ασχολείται με τα δικαιώματα των γυναικών και είναι διευθύντρια του γραφείου της Υπηρεσίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Νότιο Αφρική. Και οι δύο έχετε πέντε λεπτά. Λυπάμαι που είναι τόσο λίγο ο χρόνο μας. Καλώς ήρθατε και εσείς. Κυρία, κυρία Γέλα και κυρία Λαμίνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε. Πρόεδρε. Από την ε, Διεθνή Μνηστία είμαι και την ε, Αρμόδια Υπηρεσία του Λονδίνου, το Αρμόδιο Γραφείο του Λονδίνου. Να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή σας που μας έδωσε την ευκαιρία να απευθυνθούμε στην Επιτροπή σας σήμερα μαζί με τους συναδέλφους από τη Σουαζιλάνδη. Θα ήθελα να μιλήσω για την κρίση που υπάρχει σε ό,τι αφορά το, ε, το κράτος δικαίου, του κράτους δικαίου, την ε, ε, πρόσβαση σε ένδικα μέσα για τα θύματα των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή Βεβαίω περισσότερα θα σας πει ο α, κύριος Τζιέλη. τώρα, κάποια πράγματα για την κρίση εκεί. Είναι η δεύτερη μεγάλη κρίση κράτους δικαίου σε περίοδο μικρότερη των δεκαετών, η οποία έχει με τεράστια επίπτωση στην προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρόλο που η Σουαζιλάνδη έχει επικυρώσει πολλές από τις ε, περιφερειακές και διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ε, σύνταγμά της προβλέπει νομοθεσία ε, πολιτικών δικαιωμάτων τουλάχιστον, εξακολουθούν ε, να υπάρχουν μεγάλες, μεγάλοι περιορισμοί από την κυβέρνηση ε, των ε, δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Επίσης, Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πλήρης πρόσβαση σε κάποια ανεξάρτητη υπηρεσία για την ε, διενέργεια έρευνας για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν δείχνει να θέλει να ερευνηθούν ανεξάρτητα ε, όλα αυτά, όλες αυτές οι παραβιάσεις και οι υπεύθυνοι να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Βεβαίω πρέπει να υπάρξει λογοδοσία στην ε, δικαιοσύνη. Αυτό μέχρι στιγμή έχει γίνει μόνο μέσω των ε, δικαστηρίων και την προστασία τη ε, ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Η Amnesty International έχει εκφράσει την ανησυχία τη για την πρόσφατη διαχείριση του διαπρεπούς δικηγόρου Τόμας Μασούκου και την αφαίρεσή του από την αποχώρησή του από κάποιες δικαστικές διαδικασίες. Οι εξελίξεις αυτές ε, έγιναν ε, λίγο πριν την ακρόαση ε, της 4ης Οκτωβρίου για το UPR της Σοζηλάνδης. Δεύτερο σχόλιο για τους περιορισμούς και τις παραβιάσεις των βασικών θεμελιωδών ελευθεριών και τις ελευθερίες της έκφρασης. Αυτά τα σημαντικά πολιτικά δικαιώματα προκύπτουν μετά από δεκαετίες συγκρούσεων στη Σουαζιλάνδη. Οι επιπτώσεις των συνταγματικών διατάξεων εγγυώνται αυτά τα δικαιώματα, αλλά δυστυχώς υποσκάπτονται από κάποιες ρήτρες συγκεκριμένες περιοριστικές. Ας πούμε το, το, ότι δίνεται ε, μεγάλη σημασία στην, στο τμήμα 25 στο Σύνταγμα για την δημιουργία των πολιτικών κομμάτων. Ε, αυτό... Ε, υποσκάπτεται από το άρθρο 79, το οποίο ουσιαστικά καταργεί τη δυνατότητα ε, δημιουργίας πολιτικών, ίδρυσης πολιτικών κομμάτων. Στο, τον, στο ένα κρόαση του UPR ε, υπήρξαν κάποια ελλειπή έγγραφα για την καταχώρηση των πολιτικών κομμάτων σε, κάποιες άλλες, ε, ε, σε άλλη ακρόαση ε, ακούστηκε ότι τελικά μάλλον είναι ακόμα στα υπόψη το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν σαφής γραμμή για το τι τελικά θα γίνει. Επιπλέον, τα δικαιώματα αυτά επηρεάζονται και από καινού νόμους για τις δραστηριότητες και για την πράξη που υπάρχει για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Αυτές χρησιμοποιούνται μερικές φορές για, την, για τον περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης. Επίσης, ε, αφαίρετες ε, ε, διώξεις, συλλήψεις και με χρήση υπέρμετρης βίας από τους αξιωματούχους της κυβέρνησης χρησιμοποιούνται για να καταπιέσουν την εξάσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Και επίσης θα ήθελα πριν κλείσω να πω κάτι για τους περιορισμούς της προστασίας από του, του δικαιώματος για ενάντια της ζωής. Ε, πολλές φορές χρησιμοποιείται τεράστια βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών. Χρησιμοποιείται, χρησιμοποιούνται βασανισμοί ε, για τους συλληφθέντες. Η πρόσβαση σε ε, ιατρική βοήθεια επίσης ε, έχει περιοριστεί σε πολλές περιπτώσεις. Έχει υπάρξει λοιπόν ε, συνεπής, είναι συνεπής η θέση της κυβέρνησης ε, να μην ε, αναφερθεί στα θέματα αυτά των, της μεγάλης αμέλειας και βασανιστήριων. Υπάρχει τεράστια τιμωρησία. Μόνο μέσω του δικαστηρίου μπορεί κάποιος να ε, βρει ένα μέρος του δίκη του, παρόλο που όλη αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ αργή. Παρόλο που ε, καλωσορίζουμε την απόφαση του Πρωθυπουργού πέρσι να διερευνήσει τον ε, θάνατο ενός πολιτικού ακτιβιστή τον Μάιο του 2010, η διαδικασία αυτή απλώς τελικά δεν ε, οδήγησε πουθενά, δεν ε, δημοσιεύθηκε η έκθεση και σε ό,τι αφορά την ε, χρήση υπέρμετρης βίας για έναντι ατόμων από φτωχές κοινότητες αποτελεί άλλη μια τάση που θα πρέπει να διερευνηθεί. Τέλος, για την διάκριση κατά των γυναικών. Η συστηματική διάκριση κατά των ε, γυναικών εξακολουθεί να υπάρχει και στην νομοθεσία και στην πρακτική της Σουαζιλάνδης. Βεβαίως κάποιες αλλαγές έχουν γίνει δυνάμει του νέου συντάγματος. Οπότε δεν αποτελεί έκπληξη ότι, έκπληξη ότι εξακολουθούν να επηρεάζονται πολύ σημαντικά οι γυναίκες από την ενεργεία, την ε, επιδημία του HIV, του ιού ε, και την ανεργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. για την παρουσίαση της ε, κατάστασης στην ε, Σουαζιλάνδη. Θα ήθελα τώρα να στραφώ στους ε, προσκεκλημένους μας που έχουν συντονιστεί με την Επιτροπή μας από τη Σουαζιλάνδη. Έχετε το λόγο λοιπόν. We Περιμένετε λίγο γιατί υπάρχει ένα προβληματάκι με τεχνικό. Έχουμε τεχνικά προβλήματα. Να ακούσουμε πρώτα τον πρέσβη. Ε, όπως είπα, αντιμετωπίζουμε τεχνικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν θα θέλαμε να δώσουμε πρώτα το λόγο στον επιτετή τετραμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Σουαζιλάνδη και αν κάποιο άλλο μέλος φυσικά θα την προσωπήσετε να λάβει το λόγο μπορεί να το κάνει εδώ και στη συνέχεια θα ξαναπροσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση με τη Σουαζιλάνδη. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Yeah. Yeah. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε είμαι ο επιτετραμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σουαζιλάνδη. Λάβαμε την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας και τη διαβάσαμε προσεκτικά. Συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με αυτή την έκθεση. Συμφωνούμε στο ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας ε, του συντάγματος σε κρίσιμους τομείς. Για παράδειγμα, στο καταγραφή των ε, πολιτικών κομμάτων, η Σουαζιλάνδη παραμένει εκ των πραγμάτων μια ε, μοναρχία στην οποία ο μονάρχης έχει απόλυτες εξουσίες το σύστημα επιτρέπει συμμετοχή μόνο από άτομα και ε, όχι υπό ε, τη μορφή κόμματος και αυτό δεν βοηθάει στη δημοκρατία της χώρας. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες για την ε, κατάσταση που υπάρχει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φαίνεται να υπάρχει μια λύση, αλλά πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστούν σημαντικά ζητήματα. Συμφωνούμε ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι μάλλον οι οργανισμοί υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά λήψη ενός νόμου που θα τους το επιτρέπει. Όσον αφορά την κατάσταση των γυναικών, συμφωνούμε ότι υπάρχουν ακόμη τεράστια ελλείμματα όσον αφορά την ισότητα των φύλων ειδικότερα στον τομέα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ε, γάμου και κυδαιμονίας ε, τέκνων. Ωστόσο, παρατηρούμε κάποια σταθερή πρόοδο. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει στη σχηματισμό μιας πολιτικής για τα η ε, ισότητα των φύλων ε, που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση το νόμος ε, για τα σεξουαλικά εγκλήματα και τα εγκλήματα οικογενειακής βίας έχει ψηφιστεί και τώρα γίνεται νόμος ο νόμος για τον γάμο τώρα ακόμη βρίσκεται υπό εξέταση με χαρά ανακοινώνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα τη κατά των καταχρήσεων για βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών σε επίπεδο εκπαίδευσης, οικογένειας και κοινοτήτων. Όσον αφορά τις θεμελιώδες ελευθερίες, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες της Διεθνούς Αμνηστίας όσον αφορά τον περιορισμό της συμμετοχής πολιτικών κομμάτων και της κοινωνίας των πολιτών στην εθνική πολιτική και τη δημόσια ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο παρατηρούμε επίσης τη δυσκολία των εργαζομένων να χρησιμοποιήσουν τα μέσα ελεύθερα όπως αναφέρεται στην ε, έκθεση του ILO του 2011. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανειλημμένως έχει εξασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για τη δρακόντια νομοθεσία ασφαλείας και για τις δράσεις κατά των πολιτικών αντιφρονούντων. έχοντας όλα αυτά υπόψη. Η όλη απόδοση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σουαζιλάνδη είναι με τρίο επίπεδο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της υποσαχαρίας Αφρικής το 2010 βρισκόταν στην οικοτιστή ε, εκτιθέση από τις 53 χώρες της ε, υποσαχαρές Αφρικής. Ωστόσο αποτελεί ένα χρονισμό ύπαρξη αυτής της μοναρχίας ε, και ο, η τρόπος ζωής της βασιλικής οικογένειας είναι όλο και, θεωρείται όλο και πιο απαράδεικτη δεδομένη της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόσφατα ενέκρινε μια στρατηγική ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη Σουαζιλάνδη, κυρίω στόχο τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι να βοηθήσει τη Σουαζιλάνδη, η οποία μαζί με τη Ζιμπάμπουε παραμένει η μόνη μη δημοκρατική χώρα στην περιοχή, να εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένα δημοκρατική χώρα, όπου τα πολιτικά κόμματα θα μπορούν να δρουν ελεύθερα και όπου οι βασικέ ελευθερίε θα διασφαλίζονται και θα τις απολαμβάνουν οι πολίτες. Το ιδανικό χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι μάλλον βραχυπρόθεσμο 2013 όπου θα λάβουν χώρα οι επόμενες γενικές εκλογές. Μόνο εάν δεν μπορέσει να επιτευχθεί μέχρι εκείνη την προθεσμία, τότε θα θεωρηθεί μεσοπρόθεσμο στόχο. Ένα άλλο κύριο στόχο ε, είναι η πρόθεση τη ισότητα των φίλων σε μια κοινωνία όπου η βία κατά των γυναικών είναι ε, πολύ διαδεδομένη και όπου οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ε, περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε ιδιοκτησία. Εκτός από αυτούς τους δύο ευρύς ε, στόχους υπάρχουν και οι βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες που σχετίζονται με δράσεις κλειδιά για την πρόθεση της δημοκρατίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σουαζιλάνδη. Έχουμε την τροποποίηση της νομοθεσίας κατά της τρομοκρατίας ώστε να μην χρησιμοποιείται κατά πολιτικών ακτιβιστών για την απαγόρευση ε, πολιτικών κομμάτων και πολιτικών δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Δημόσιας Διοίκησης σε ένα πλήρως λειτουργικό σώμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη. Με ενημερώνουν ότι λύθηκαν τα τεχνικά προβλήματα τώρα.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 Δυστυχώς δεν ακούγεται. Οι διερμηνείς δεν μπορούν να μεταφράσουν, δεν ακούγεται αρκετά η φωνή για να καταλάβουμε τι λέει ο μιλητής από το βίντεο.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 συνεχίζει πολωνικά ο πρόεδρος. Παρά τις τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, μπορέσαμε παρόλα αυτά να ακούσουμε ε, στα αγγλικά τους μιλητές, οι οποίοι παρόλο που μίλησαν πάνω από τα λεπτά που τους είχα διαθέσει, μας είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και βλέπουμε ότι τελικά τα ίδια προβλήματα εμφανίζονται παντού, όπου έχουμε να κάνουμε με συνταγματικά ζητήματα, ε, θέματα δικαιοσύνης θέματα που έχουν να κάνουν με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα θέλω να αρχίσουμε τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, πως κάποιος ευρωβουλευτής θέλει το λόγο, παρακαλώ κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία να μπει στην ημερήσια διαταξή μα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σουαζιλάνδη. Και ευχαριστώ και τους φίλους που μας μίλησαν από την Σουαζιλάνδη. Όπως είπατε, πράγματι, μας έδωσαν την εικόνα που είναι ίδια κάθε φορά όταν έχουμε να κάνουμε με την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στον νόμο και στην πράξη. Βέβαια στις χώρες μας ε, δεν είναι ακριβώς ε, τα ίδια. Από ό,τι φαίνεται ε, στην χώρα τους, από ό,τι μας περιέγραψαν, τα πράγματα είναι πιο σοβαρά και πιο συστηματικές οι παραβιάσεις. Και η απόσταση είναι μεγαλύτερη ανάμεσα στον νόμο και στην πράξη. Ανάμεσα στο κράτος δικαίου και τις διακρίσεις που γίνονται σε βάρος των γυναικών. Διακρίσεις που είναι πολύ συνηθισμένες. Όμως και πριν έχω ακούσει τους φίλους μας και τον κύριο Ρέινα, κοιτώντας το κείμενο της υπουργικής απάντησης στο UPR από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στα συνταγματικές υποθέσει της Σουαζιλάνδης, έχω την αίσθηση ότι κάτι άσχημο υπάρχει εδώ. Και κάτι χοντροειδές θα έλεγα και ορισμένα κεφάλαια. Και ιδιαίτερα σχετικά με το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τις γυναίκες και τα πολιτικά τους δικαιώματα. Γιατί τελικά τι νόημα έχει στο Σύνταγμα σε κάποιο άρθρο να λέει ότι ναι, έχουν πολιτικά δικαιώματα κτλ. Και, και σε ένα άλλο άρθρο να εμποδίζονται από το να είναι υποψήφιες στις γενικές εκλογές. Επειδή, λέει το άρθρο αυτό, οι υποψήφοι πρέπει να εκλέγονται βάσει των προσωπικών της προπτικής τους αξίας. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, χωρίς πολιτικά κόμματα, μα είναι, είναι αστείο, είναι γελίο, σχετικό κορυδία. Έπειτα, οι γυναίκες από τις πληροφορίες που ακούσαμε, αλλά και από άλλες πηγές, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και επιδεινώνεται ε, με το AIDS, που βέβαια οι γυναίκες είναι κατά κύριο λόγο διπλά θύματα. Ένα άλλο σημείο που, στο οποίο, το οποίο πρόσεξε όλους ιδιαίτερος από την απάντηση εδώ είναι που λέει ότι δεν είναι υποχρεωτική η θανατική ποινή. Χα, χα. Και λέει ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες, κάποια ελαφρυντικά και καταλήγει στο ότι η Σουαζιλάνδη ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται η θανατική ποινή από το 1983 και ότι άρα θεωρείται ότι έχει καταργήσει τη θανατική ποινή. Μα όλα αυτά εμένα με βάζουν σε σκέψεις γιατί υπάρχει ατιμορρησία τελικά στη Σοζιλάνδη και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι πολύ πιο έντονες όσον αφορά τις αντιδράσεις τους απέναντι στην Σουαζιλάνδη και να ζητήσουν από τη Σουαζιλάνδη να κάνουν αυτά για τα οποία έχουν δεσμευτεί. Να φέρουν σε πέρας όλες τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα μετά την κυρία Γκόμες. Πρέπει να πω ότι ο πρέσβης Τζονέκο είναι εδώ στην αίθουσα και γι' αυτό θέλω να το ρωτήσω, μήπως θέλετε το λόγο, κύριε Πρέσβη, Ζωέλ Λεκό. Εφόσον ε, επιθυμείτε, παρακαλώ σε πέντε λεπτά να μας δώσετε τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ελληνική σας πρόσκληση σε αυτή τη συνεδρίαση και Παρακαλώ να έχετε κατανόηση αν δεν ανταποκριθούμε στις ε, προσδοκίες σας. Επειδή αυτή είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο φόρουμ, εμείς ως πρεσβεία του Βασιλισσίου του Σουαζιλάνδης ε, εκτιμούμε αυτή την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σουαζιλάνδη, ειδικότερα τα δικαιώματα των γυναικών. Κύριε Πρόεδρε, επειδή μόλις πριν από ένα μήνα η κυβέρνηση της ε, Σουαζιλάνδης ε, ε, παρουσίασε την εθνική έκθεση για τα ανθρωπιστικά δικαιώματα στην Σουαζιλάνδη στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΠΑ στη Γενέβη. Ελπίζουμε Ελπίζουμε ότι η εκθέσή μας ε, απέδειξε τις προσπάθειες που κάνουμε για την ε, υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου που μίλησε πριν από μένα αναφέρθηκε στην ε, ομιλία αυτή του Υπουργού Πιστεύω ότι και το δώσω ολοκληρωτικά τη δήλωση και τις ε, απαντήσεις που έδωσε η κυβέρνηση εκείνη την ημέρα, είμαι βέβαιος ότι θα εκτιμήσετε το γεγονός ότι η Σουαζιλανδή έχει δεσμευτεί στη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προφανώς η χώρα μου έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Προσδοκία μας σήμερα είναι πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί μια ευκαιρία να μοιραστούμε τις πρακτικές μας και να βελτιωθούμε περαιτέρω μέσω επικοδομητικού και αντικειμενικού διαλόγου με τους εταίρους μας, ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή λοιπόν μας σήμερα εδώ περιορίζεται στο να ακούσουμε τις απόψεις των αξιοτιμών μελών αλλά θα ήθελα να απαντήσω με τη θέση της κυβέρνησής μου. Η Σουαζιλάνδη έχει δεσμευτεί ώστε να διασφαλίσει ε, το πλήρε φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το λαό τη, όπω προβλέπεται στο Σύνταγμα, παρά τι οικονομικέ προκλήσει που αντιμετωπίζει. Καθώ μιλάμε σήμερα, η Σουαζιλάνδη αντιμετωπίζει σήμερα μία δυσμενή οικονομική κρίση που θέτει πολλούς φραγμούς ε, και πολλά προβλήματα σε όλες τις λειτουργίες της κυβέρνησης, ακόμη και στις προσπάθειες βελτίωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. οι ελλείψει ε, στις προσπάθειε αυτές βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οφείλονται σε ελλείψει ε, δυνατοτήτων, δυναμικού. Και γι' αυτό τον λόγο ο Υπουργό, όταν παρουσίασε τη δήλωσή του είπε ότι εμείς ως χώρα με την υποστήριξη, χρειαζόμαστε υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα ώστε να δώσουμε ε, δυνατότητα στους οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων να οικοδομήσουν δυνατότητα για την ανάπτυξη μια στρατηγικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενός σχεδίου δράσης στην εντατικοποίηση της ευαισθητοποίησης του γενικότερου κοινού και όλων των ενδιαφερομένων. Υποστηρίζοντας την ευθυγράμμιση των εθνικών νόμων με τη Διεθνή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Σύνταγμα. Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας ε, τις παρατηρήσεις των εδωμελών και των συμπατριωτών μου όλες οι δηλώσεις που ακούσαμε επικεντρώνονται στο γεγονό ότι η Σουαζιλάνδη δεν έχει τη δυνατότητα. Αυτό καταδεικνύουν όλες αυτές οι δηλώσεις. Δεν έχει τη δυναμικότητα που, που να επιτρέπει ότι θα διασφαλιστεί ότι θα υλοποιείται ο νόμος ε, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά συνέπεια εμείς ως κυβέρνηση κύριε Πρόεδρε εκτιμούμε ιδιαίτερα την ε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βασίλειο της Σουαζιλάνδης υποστηρίζει τη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους, ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε διατεθειμένοι να ξεκινήσουμε διάλογο μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, με αυτές τις λίγες παρατηρήσεις μου επαναλαμβάνω ξανά το γεγονός ότι οι δηλώσεις του Υπουργού και όλες οι εκθέσεις Τις επικροτούμε, τις υποστηρίζουμε και ελπίζουμε ότι όλα τα μέλη θα εξετάσουν αυτά τα ζητήματα υπό αυτό το πρίσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη, κυρίες και κύριοι. Αυτή η δήλωση του κυρίου Πρέσβη μου φαίνεται εξαιρετικά σημαντική ακούγοντας τον ε, κοιτούσα την αντίδραση των προσκεκλημένων μας στην οθόνη οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στη ε, συζήτησή μας μέσω της ε, σύνδεσης μέσω διαδικτύου από τις εκφράσεις των πρόσωπά τους καταλαβαίνω ότι δεν συμφωνούσαν σε όλες τις περιπτώσεις πιστεύω ότι αυτό θα αποτελεί στην αρχή ενός διαλόγου που θα χρειαστεί να λάβει χώρα η Επιτροπή μας ε, είναι καλό που συμμετέχει στη γέννηση αυτού του διαλόγου. Θα ήθελα αυτή η συζήτηση γιατί ο Σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Σουαζιλάνδη να φέρει αποτελέσματα μακροπρόθεσμα όταν εξετάζουμε την Εθνική Στρατηγική της Σουαζιλάνδη που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι προβλέπονται ελάχιστε θέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα παρότι αυτό αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της πολιτικής μας. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό επειδή πριν λιγότερο από μία ώρα συζητούσαμε για την νέα στρατηγική ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε στον τομέα των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βαζιλάνδης. Είμαι πεπισμένος ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τις αρχές της Σουαζιλάνδης ώστε να προβούν σε μεταρρυθμίσεις ακόμη πιο βαθιές. Παρότι έχουν γίνει ήδη ορισμένες αλλαγές όπως είπε ο κύριος Πρέσβης όπως υπογράμμισε επίσης και ο, ο πρέσβης της ε, αντιπροσωπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευχαριστώ την κυρία Ρένερ Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους από τη Σουαζιλάνδη που είχαν την υπομονή να αναμένουν ε, την αποκατάσταση της σύνδεσης μετά τα τεχνικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν κλείνω αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και περνάμε στο επόμενο. Θα ήθελα λοιπόν να παράσω στην ανταλλαγή απόψεων με τον Κριστιαν Έλερ, πρόεδρο της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο σχετικά με την επίσκεψη της Αντιπροσωπείας στη Βόρεια και Νότια Κορέα που έλαβε χώρα από 28 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου 2011. Τα μέλη αυτής της Αντιπροσωπείας είχαν την ευκαιρία να μεταβούν σε αυτές τις δύο χώρες ε, στο πλαίσιο της διακοινοβουλευτικής συνάντησης μεταξύ της Ένωσης και των Διευθών χωρών. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επικεντρώνεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα. Θυμόμαστε τις συνεδρίες που είχαμε διοργανώσει τον Απρίλιο του 2010. Εκεί ακούσαμε τον κύριο Τσίγκοντζο ο οποίος ε, διέφυγε από ένα στρατόπεδο κράτηση της Βορειας Κορέας. Ακούσαμε επίσης τη μαρτυρία του αντιπροσώπου για το ζήτημα της Βορειας Κορέας ε, στο Υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Ιούλιο 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα για, στη Βόρεια Κορέα. Ξεκίνησε μία ερευνητική επιτροπή και με κριτική στις αρχές για τη συστηματική και σοβαρή παραβίαση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Η Προεδρία της ε, Επιτροπής μας, ε, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις επισκέψεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ζήτησε από τα μέλη της αντιπροσωπείας να προσέξουν ιδιαίτερα ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βορεια Κορέα. Ο κ. Κρίστιαν Ελέρε, πρόεδρος της αντιπροσωπείας, θα μοιραστεί μαζί μας τις εντυπωσει που σχημάτισε. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Έλερ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα μιλήσω γερμανικά. Καταρχάς να ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των αντιπροσωπιών και της Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό μετά τη Λισαβόνα το Κοινοβούλιο να εμπλέκεται σε τέτοια θέματα και εξειδικευμένα αλλά και γενικά όπως τα θέματα εξωτερικά αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συνεργασία λοιπόν μεταξύ των Επιτροπών είναι πολύ σημαντική καθώς επίσης και η συνεργασία με την, υπηρεσία, με την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Τώρα, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ με τις ε, ε, λεπτομέρειες. Ήταν η τρίτη προσπάθεια που κάναμε να πάμε στη Βορεια Κορέα. Οι δύο πρώτες ε, απόπειρες είχαν καταρρεύσει γιατί υπήρξαν πολλές προβοκατόρικες κινήσεις στα σύνορα, υπήρξε, υπήρξαν κάποιοι κάποιες αντιδράσεις στα σύνορα. Είχαμε ακυρώσει λοιπόν κάποιες από τις, ε, τη μία από τις δύο ε, επισκέψεις. Τώρα ήταν η τρίτη φορά που προσπαθήσαμε να πάμε. Σε κάθε ταξίδι που κάνει η αντιπροσωπεία προσπάθησε με τον σωστό τρόπο και διπλωματικά να θίξει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε πόσο δύσκολο θέμα είναι αυτό. Ποτέ δεν λαμβάνει κανείς μια ευθεία απάντηση από την Βόρεια Κορέα. Απλώς έτσι διατισταθλασμένης μας απαντούν για το πόσο είναι έτσι, έτοιμοι να μπουν σε ένα διάλογο. Το σημαντικό, κατά την άποψή μας, είναι ότι είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα στη χώρα, επιτόπου. Το θέμα των ανθρωπινών δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα συνδέεται άρρηκτα με το θέμα της, των συνθήκων διαβίωσης των ε, πολιτών και της παροχής τροφίμων στην Βόρεια Κορέα. Ε, είχαμε λοιπόν, ε, το, είδαμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. τώρα βέβαια αυτή είναι δική μου εντύπωση αλλά στην Βόρεια Κορέα τώρα είναι, οι εισοδιές είναι πάρα πολύ λίγες, αλλά βρίσκονται στα, στα χωράφια και βλέπετε παντού α, τις οδιές, όλα ο, βλέπετε παντού να αναγράφεται ότι λόγω του ότι πρόκειται να είναι 100, θα γιορταστούν τα 100 χρόνια της ε, ε, επαιτίου της ε, ανάληψης της κυβέρνησης από τον Κιμ jong και παντού υπάρχουν πινακίδες που λένε ότι εκείνη την ημέρα των εορτασμών οι Βορειοκορεάτες δέχονται να φάνε μόνο δύο φορές και το ένα τους γεύμα να το παραχωρήσουν στον, στον, για τους εορτασμούς της επαιτίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλος καταναγκασμός είναι αυτός, ακόμη και για τα βασικά όπως είναι τα τρόφιμα. Είναι λοιπόν μια χώρα που είναι πολύ ιδιαίτερη. Η κατάσταση τώρα η επιστηστική στην χώρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το καθεστώς ακριβώς λόγω των εορτασμών τον επόμενο χρόνο ήδη προσπαθεί να δημιουργήσει αποθέματα έτσι ώστε του χρόνου που θα γίνει ο εορτασμός να έχει έτσι ένα, να, να μπορεί να παρουσιάσει μια ε, αντιπροσωπευτική εικόνα του ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παροχή τροφίμων παρόλο που αυτό δεν είναι αλήθεια γιατί τα πράγματα είναι τελείως αντίθετα. Είναι ε, έτσι, επέμβαση στη ζωή των, των πολιτών δραματική. Ε, αυτοί που τους ζητείτε να απόσχουν από το ένα γεύμα, μόνο και μόνο για να μπει η ποσότητα αυτή στο απόθεμα για τους εορτασμούς. Επίσης, κάναμε κάποιες συζητήσεις και με τον ύπατο εκπρόσωπο και με τους, ε, συν, με τους φίλους από την, νότια, από την Νότια Κορέα συζητήσαμε το θέμα του, του τι θα γίνει με την κυρία Σιν. Ξέρω ότι είναι πολλές οι λυπηρές ιστορίες σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες και μπορεί να αναρωτιέστε γιατί ασχοληθήκαμε με αυτό το πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά τώρα το θέμα είναι αν η Βόρειος Κορέα είναι διατεθειμένη να δώσει μέσω έστω ενός παραδείγματος ένα σωστό μήνυμα. Γι' αυτό λοιπόν προχωρήσαμε λίγο παραπάνω. Θέσαμε λοιπόν τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μιλήσαμε για συγκεκριμένες αποφάσεις σε σχέση με, την, ε, ε, με τα υποστηρικτικά προγράμματα για την παραγωγή τροφίμων. Μιλήσαμε για το ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα μήνυμα από την αντιπροσωπεία της Βορειού Κορέας εδώ στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι γενικώ το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Βόρειο Κορέα δεν οδηγεί ποτέ σε απάντηση. Οπότε πρέπει και εμείς να είμαστε λίγο πιο αυστηροί. Ίσως ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχουν, ε, υπάρχει κάποια μετακίνηση από τις άτεκτες θέσεις του στη μία ή την άλλη περίπτωση. Επίσης, ενίσχυση των, ε, του επιστημιστικού προγράμματος, η υποστήριξη της παραγωγής, η δομικά δηλαδή, η δομική υποστήριξη της παραγωγής, να δούμε αν υπάρχει μετακίνηση στον τομέα αυτό και σε ποιο βαθμό η Βόρειος Κορέα είναι διατεθειμένη να μπει σε έναν διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή λοιπόν είναι η δική μου πρόταση. Ξέρω ότι η Επιτροπή σας σκέφτεται να υποβάλει ένα ψήφισμα. Ναι, να είναι έτσι αρκετά γενικόλογο, αλλά να συνδεθεί και με συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι σαφές το ότι ο τρόπος της συμπεριφοράς της χώρας, η κλειστοφοβική έτσι, ε, ατμόσφαιρα που επικρατεί στην χώρα θα δυσκολέψει βεβαίως πολύ την αλλαγή της κατάστασης και της νοοτροπίας. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Υπάρχουν κάποιε ε, μεμονωμένες περιπτώσεις. Ας ζητήσουμε λοιπόν μέσω αυτών των μεμονωμένων περιπτώσεων από τη Βόρεια Κορέα να κάνει ένα βήμα προς τα μπρος και να στείλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν μπορούμε και από εδώ, από τις Βρυξέλλες, να, να, να δώσουμε ένα, ένα μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα... Ήθελα λοιπόν να σας αναφέρω και κάποια πράγματα και για τους πολιτικούς κρατούμενους. Πήγαμε σε, ένα από τα προγράμματα και βρήκαμε, έτσι μια, βρήκαμε μια ηλικιωμένη κυρία που, μας, που τη ρωτήσαμε πώς να πάμε στο, στο πρόγραμμα αυτό. Δεν μπορούσε να μας απαντήσει. Και ένας από τους αξιωματούχους εκεί τη ζήτησε να ξαπλώσει στο, στο χώμα με το πρόσωπο προς τα κάτω γιατί ήθελε έτσι να την ε, εξευτελίσει γιατί δεν μπορούσε να μας δώσει τις πληροφορίες που θέλαμε, να μας δείξει το δρόμο. Επίσης, έπρεπε να είναι με το πρόσωπο αυτή η γυναίκα στο, στο χώμα. Να, δηλαδή, φανταστείτε πόσο ε, υποτιμητικό είναι αυτό για την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου. Μια ηλικιωμένη γυναίκα τώρα να είναι εξαπλωμένη με το πρόσωπο στο χώμα επειδή δεν ήξερε να μας δείξει το δρόμο. Βεβαίως, ε, μετά εμείς προχωρήσαμε ε, υποθέτω ότι η γυναίκα αυτή δεν σηκώθηκε αμέσω. Ε, είναι τόσο δηλαδή η υποτέλεια κάποιων ε, μερικέ φορέ ε, στην οποία υποχρεώνονται οι άνθρωποι, που πραγματικά ήταν συγκλονιστικό που το είδαμε. Εμένα ο πατέρας μου ήταν πολιτικός κρατούμενος στην Γερμανία. Δεν έχω δει καμία άλλη χώρα που να έχει τόσο μεγάλη επέμβαση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων όπως η Βόρεια Κορέα. Ας πούμε, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάντα έχει να κάνει με την τροφή, με κάποια έτσι ανθρώπινα βασικά δικαιώματα. Για παράδειγμα, ε, κόβεται το ρεύμα και η παροχή ενέργειας ως πολιτικό ε, μέσο επιβολής. Ε, κόβεται το ρεύμα σε συγκεκριμένους δρόμους, σε συγκεκριμένα τετράγωνα. Ε, αυτά τα πράγματα προφανώς πιέζουν πολύ την ε, ε, καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Γιατί ουσιαστικά είναι μια, ένα είδος ομοιρίας μιας ολόκληρης, ενός ολόκληρου Βεβαίω οι δυνατότητε που έχουμε για να, δυνατότητες που είχαμε να έρθουμε σε επαφή με, την, ε, με τους οπλούς πολίτες ήταν πολύ περιορισμένες, ε, οπότε πρέπει να δούμε τώρα αν αυτό έχει σχέση και με, τις, με τους εορτασμούς του επόμενου έτους, αν δηλαδή θέλει κανείς να δημιουργήσει μια εικόνα προς τα έξω ε, και θέλει να διακόψει πούμε αυτή την ε, εντύπωση που υπάρχει για πολιτική απομόνωση. Προσπαθήσαμε να επισκεφθούμε λοιπόν ε, αρκετά σημεία στην ε, Pyongyang. Υπάρχουν ε, βεβαίως και πολλές ιδιωτικές έτσι, αγορές. Τώρα φανταστείτε γυναίκες που κάθονται με ένα φακό τη νύχτα και πουλάνε το, τα προϊόντα τους. Κάτι τέτοιο είναι οι ιδιωτικές αγορές στην Βόρειο Κορέα. Και μάλιστα ένα κιλό ντομάτες μπορεί να σημαίνει τρεις φορές το μηνιαίο μισθό ενός ε, πολίτη. Οπότε το θέμα εδώ είναι ότι υπάρχει μεγάλη ε, διαστρωμάτωση στην ε, Βόρειο Κορέα και το θέμα της παροχής ε, προνομίων, αν μπορούμε να πούμε ότι η παροχή τροφής είναι ένα προνόμιο, είναι πάρα πολύ ε, συγκεκριμένη. Αυτό μπορεί να συνέβαινε, ας πούμε, στην Ευρώπη τον 17ο αιώνα όταν υπήρχαν ε, ε, σε μικρά χωριά κάπου στην Ευρώπη συλλογικές ε, συνεταιριστικές παρεμβάσεις για την παροχή ενέργειας, για την παροχή τροφίμων κτλ. Υπάρχει λοιπόν έτσι μια συλλογική ποινικοποίηση των πολιτών στη Βόρειο Κορέα που ουσιαστικά είναι και αυτό ένα μέτρο καταπίεσης. Ένα άλλο παράδειγμα. Ε, ένα, ένα σπίτι πρέπει να έχει σε κάθε ε, δωμάτιο ε, έναν τοίχο ελεύθερο για εικόνες των ηγετών του. Αν το σπίτι καεί, η υποχρέωση των ανθρώπων αυτών είναι να σώσουν τις εικόνες. Γιατί αλλιώς ε, έχουν να πληρώσουν, ε, τους επιβάλλονται μεγάλες ε, ποινέ. Δεν μιλούμε δηλαδή για τα υπάρχοντα του σπιτιού, μιλούμε για τη διάσωση της εικόνας του ηγέτη της χώρας, αν το σπίτι τους καεί. Και μια τελευταία πρόταση. είναι με μονομένα βεβαίω τα παραδείγματα αυτά, αλλά είναι έτσι μια γενική εικόνα που επικρατεί. Εμείς προσπαθούμε στα πλαίσια του διαλόγου. Νομίζω όμως ότι σκόπιμο θα ήταν να έχουμε μια τέτοια δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το, κράτος, από το Κοινοβούλιο και να χρησιμοποιηθεί αυτό το 2012 γιατί θα αποτελέσει ένα έτος σύμβολο αυτό για την Βόρεια Κορέα. Και καλό θα ήταν ο εισηγητής, εμείς ήρθαμε σε επαφή με τον εισηγητή μάλιστα. Ο ε, εισηγητής λοιπόν από την ε, Επιτροπή στο Α να είναι ίσως ε, να, συμμετάσχει. Ε, νομίζω ότι είναι σωστό να γίνουν οι απαραίτητες ανταλλαγές απόψεων, πληροφοριών ε, μεταξύ της ΣΤΟΑ και της ε, Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εγώ ευχαριστώ κύριε Έλερ. Ε, πολύ πραγματικά, πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Είναι πραγματικά τρελή η κατάσταση που επικρατεί εκεί. Είναι απίστευτη. Τώρα θα ήθελα να καλέσω να πάρει το λόγο ο κύριος Μπραντς. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σχετικά σύντομος. Ανησυχούμε σοβαρά για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βόρειο Κορέα. Μας ανισχύει η χρήση βασανιστήριων, η ύπαρξη στρατοπέδων εργασίας, η εκτενής χρήση της θανατικής πύρνης, οι σοβαροί περιορισμοί της ελευθερίας σκέψης, έκφρασης, συνάθρησης και θρησκευτική θρησκευτικών πεπιθήσεων καθώς και ο πλήρης αποκλεισμός του πληθυσμού από οποιοδήποτε είδους δημόσιες υποθέσεις. Επίσης μας ανησυχεί η ανθρωπιστική κατάσταση και η επισητιστική κατάσταση στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος ε, Χέλλερ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει προσπάθειες, είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε κάτι για όλα αυτά οι προσπάθειές μας αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης σε διεθνές επίπεδο και σε κάποιες διμερείς επαφές που έχουμε σε διεθνές επίπεδο. Δραστηριοποιούμαστε κυρίως στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενική Συνέλευση την περασμένη εβδομάδα των Ηνωμένων Εθνών εγκρίθηκε πάλι ένα ψήφισμα το οποίο παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταδικάζει την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βόρεια Κορέα. Αυτό το ψήφισμα εγκριθήκε για έκτη φορά. Έκτη φορά ε, παρουσιάζουμε ένα τέτοιο ψήφισμα. Εγκρίθηκε με ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία από την πέρυσι. 112 κράτη ψήφισαν υπέρ αυτού του ψηφίσματος. Επίσης υποστηρίζουμε τον ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών που ορίστηκε από το 2004 και πιεζούμε τις αρχές της Βορειας Κορέας να παρέχουν πρόσβαση σε αυτό τον εισηγητή στη χώρα. Επίσης πιεζούμε τις αρχές της Βορειας Κορέας να λάβουν υπόψη τις ε, συστάσεις ε, που έγιναν στο UPR, στο Συμβουλίο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων στη Γενέβη το 2009 η Νότια Κορέα, η Βόρεια Κορέα απλά αρνήθηκε, απέρριψε όλες αυτές τις συστάσεις σε διμερές επίπεδο, ετησίως, ε, διεξάγεται πολιτικός διάλογος με τη Βόρεια Κορέα. Τονίζουμε τη σημασία της συνέχισης των διμερών, ε, του διμερούς διαλόγου για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αρχές του 2000 Τις δεκαετές του 2000 είχαμε διμερή διάλογο με τη Βόρεια Κορέα αλλά όταν αναλάβουμε την πρωτοβουλία στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών οι, Βόρει... οι αρχές της Βόρειας Κορέας ένιωσαν προδομένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διέκοψαν το διάλογο το διμερή διάλογο επίσης τακτικά συζητάμε με τους Κινέζους ε, για το θέμα της Βόρειας Κορέας και των προσφύγων, αλλά εκεί να αρνείται λεπτομερή συζήτηση για αυτό το ζήτημα, ισχυριζόμενοι απλά ότι οι πρόσφυγες ε, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με, το διεθνή, με τη διεθνή νομοθεσία. Ορισμένα από τα σημεία που ανέφερε ο κ. Χέλλερ η, η κατάσταση, θα σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε τον Ιούλιο να παρέχει υποστήριξη 10 εκατομμυρίων για επιστημιστική παροχή στο WFP. Το ζήτημα πολιτικής εκπροσώψης της Βόρειας Κορέας εδώ. Έχουμε πολιτικές σχέσεις εδώ και 10 χρόνια, αλλά δεν έχουμε ανταλλαγή ε, πρεσβειών. Έχουμε εξηγήσει στη Βόρεια Κορέα για να, ότι για να έχουμε μια τέτοια ανταλλαγή να υπάρχουν πρέσβεις θα πρέπει να δούμε προόδο για το ζήτημα των πυρηνικών που αποτελεί και το μείζον ζήτημα με τη Βορειοκορία αλλά φυσικά υπάρχει και το ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Κύριε Γκόμες. In the late 80s and at that time there was... Στα τέλη της δεκαετίας του 80 ήμουν εκεί και τότε συζητούσαμε πολύ για Ιαπωνέζους που είχαν απαχθεί από την Βόρεια Κορέα ώστε να χρησιμοποιηθούν ως κατάσκοποι, ξέρω εγώ τι. Τότε που τα είχα ακούσει αυτά, έλεγα «Α, αυτά είναι προπαγάνδα των Ιαπώνων». Αλλά μετά από μερικά χρόνια αναγκάστηκα να το πιστέψω, γιατί επιβεβαιώθηκε από τις ίδιες τις αρχές της ε, Βόρειας Κορέας ότι είχαν απάγει τους ε, Ιαπωνέζους αυτούς για να τους χρησιμοποιήσουν είτε για να διδάξουν Ιαπωνικά είτε ως κατασκόπους και άλλα τέτοια. Μα είναι μια παράλογη, ένα παράλογο καθεστώς, ένα τρελό, εκτός λογικής. Άκουσα τις ιστορίες του κύριου Έλερ με την γυραιά αυτή κυρία. Μα πραγματικά είναι ταπεινωτικό. Αυτό το καθεστώς δεν έχει... Δεν το διαφέρει ούτε στο ελάχιστο η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν διαφωνώ με το γεγονός ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσα έχουμε για να υπάρχει κάποιος διάλογος, να ρωτάμε αυτά που θέλουμε να ρωτήσουμε κτλ. κτλ. Αλλά το καθεστώς αυτό δεν θα μπορούσε να κρατηθεί στην εξουσία αν δεν το στήριζε το κινέζικο καθεστώς. Φυσικά έχουν και αυτοί τα δικά τους τα προβλήματα, αλλά καμία σχέση με τη στάση της Βόρειας Κορέας. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το ζήτημα αυτό να το συζητήσουμε πολύ περισσότερο με τους Κινέζους. Ξέρω ότι στο τελευταίο μας ψήφισμα το λέμε αυτό. Και άκουσα και αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που τόνισε ε, ότι οι Κινέζοι αποφεύγουν το θέμα είναι δυνατόν να του επιτρέπουμε να αποφεύγουν το θέμα, γιατί οι Κινέζοι είναι οι γείτονε τη Βόρειας Κορέας που συντηρεί το καθεστώς αυτό. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν οι Κινέζοι να συνεχίζουν να στηρίζουν ένα τέτοιο καθεστώς. Πρέπει να το θέσουμε σε αυτούς με μεγαλύτερη ισχύ στο διάλογο που έχουμε με την Κίνα αλλά και με τον κόσμο, με το κοινό. Στην Κίνα να συζητήσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Γκόμες, τώρα ο κύριος Έλερ ίσως για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Όντως, εγώ έζησα αυτή την εμπειρία η αντιπροσωπεία ουσιαστικά τι προτείνει. Προτείνει να συνεχίσουμε με αυτόν τον μερικές φορές παράλογο διάλογο. Όμως νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό με μικρές δόσεις. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Γίνονται πολλές συζητήσεις για επισητιστική βοήθεια. Επισητιστική βοήθεια που είναι ένα μη πολιτικό πρόγραμμα. Άρα δεν θα μπορούσαμε εδώ να βάλουμε όρους, προϋποθέσεις για να το θέσουμε σε εφαρμογή. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια ελιγμών. Δηλαδή η επιχειρηματολογία της ε, ΕΚΟ δεν έχει να κάνει με ολόκληρη την κατάσταση. Ξέρουμε ότι η έκκληση για επιστηστική βοήθεια ήταν ένας πολιτικός ελιγμός για να αποφευχθεί η πολιτική απομόνωση. Γιατί όταν ζητάει κάποιο ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορείς να αρνηθείς να συζητήσεις. Άρα έτσι διακόπτεται ο διπλωματικός αποκλεισμός. Ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση αυτή από την Βόρεια Κορέα να ζητήσει επισητιστική βοήθεια. Γιατί τότε αναγκάζονται όλοι, εφόσον δεν πρόκειται για πολιτικό θέμα εξορισμού, αναγκάζονται όλοι να μπουν σε αυτό το διάλογο. Η επιχειρηματολογία λοιπόν της ΕΚΟ υπέρ της επιστημιστικής βοήθειας δεν αφορά την ε, όλη κατάσταση, αφορά ορισμένες κατηγορίες ε, άτομα με αναπηρίες κλπ. Ξέρουμε ότι η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε κάλλιστα να βλύνει το πρόβλημα. Αλλά υπάρχει καταρχήν το πρόγραμμα για το στρατό, οι οποίοι μαζεύουν τρόφιμα για να έχουν την επόμενη χρονιά. Αν λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να κάνει κάτι, θα μπορούσε να διατυπώσει κάτι που να μην είναι μεν μια πολιτική προϋπόθεση, πολιτικός όρος, αλλά να έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να είναι ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι πρέπει τα τρόφιμα αυτά να είναι για τους ανάπηρους. Να ζητάμε, αν μη τι άλλο, να επικυρώσει τη σύμβαση για τα άτομα με αναπηρία στη Βόρεια Κορέα. Είναι δηλαδή ένας πλάγιος τρόπος, ένας έμεσος τρόπος να ζητήσουμε η επιστηστική βοήθεια να πάει και στα άτομα με αναπηρίες. Νομίζω ότι τουλάχιστον, αν μη τι άλλο στην επιχειρηματολογία μας, πρέπει να το προσθέσουμε αυτό, ότι αν θέλουμε επιστηστική βοήθεια ε, να πηγαίνει και στα άτομα με αναπηρίες, το καθεστώς εκεί πρέπει να το κάνει. Βέβαια είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί εμείς προσφέρουμε κάτι που δεν είναι πολιτικό, οπότε πώς μπορείς να συνδέσει ένα πολιτικό θέμα με την βοήθεια αυτή. Και απ' την άλλη δεν πρέπει να το βγάζουμε από το μυαλό μας, άρα πρέπει να βρεθεί μια διάμεση λύση. Για παράδειγμα, η σύμβαση αυτή των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα αν επικύρωναν τη σύμβαση αυτή. Και γιατί στη Βόρεια Κορέα δεν βλέπεις άτομα με αναπηρίες, δεν τους βλέπεις. Και κάποιοι συνάδελφοι το έθεσαν. Πού βρίσκονται αυτοί. Και οι απαντήσεις που μπορείς να φανταστείς είναι φρικεστικέ βέβαια. Από το τίποτα μέχρι διάφορα που μας τρομάζουν. Και έχω και εμπειρίες από κάποια κράτη-μέλη στο παρελθόν, κάτω από συγκεκριμένα καθεστώτα, όπου τα άτομα με αναπηρίες εξαφανίζονταν με φρικτό τρόπο. Και υπάρχουν στην Ευρώπη τέτοιες εμπειρίες από το παρελθόν όσον αφορά τη συμπεριφορά απέναντι στα άτομα με αναπηρίε. Και το ίδιο φοβόμαστε και για τη Βόρεια Κορέα. Προφανώ και υπάρχουν άτομα με αναπηρίε, τα οποία όμω δεν ανταποκρίνονται στο ιδεώδε που έχει το καθεστώ για την ε, κοινωνία του. Και άρα δεν πρέπει να εμφανίζονται. Θα φτάσουμε στο τέλος στο σημείο που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά, αλλά μη τι άλλο, κάθε βήμα που κάνουμε υπέρ της επιστηστικής βοήθειας να συνδέεται με κάποιο τρόπο να αποτελεί ένα έστω μικρό βήμα όπως ε, αυτό που είναι για την επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων ε, Εθνών για τα άτομα αναπηρίας, που δεν είναι πολιτική κίνηση αυτή καθ' αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Λέρ. ποιο καθεστώς αυτού του είδους σέβεται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όχι, ο κύριος Σέλλερ με αυτά που μας είπε μας το αποδεικνύει αυτό κατάφορα. Κάποιοι στη Βόρεια Κορέα, ε, σύμφωνα με το καθεστώς εκεί, δεν αξίζουν το ίδιο όπως και οι υπόλοιποι να αντικρίζουν το φως της ημέρας κάθε μέρα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η ιστορία αυτή για την ε, ε, μεγάλη γιορτή που έχουν του χρόνου είναι μια ευκαιρία η χώρα αυτή να δείξει τη δύναμή της. Είναι θλιβερό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις πρώτες εντυπώσεις που είχα από τις αλλαγές στην Αλβανία. Είχα πάει τότε στη χώρα και όταν το αεροπλάνο μου πλησίαζε στο αεροδρόμιο στα Τύρανα, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η θέα καταφυγίων. Πάρα πολλά που φτάνανε μέχρι την ακτή, που είναι και μια υπέροχη ακτή εκεί στην Αλβανία, αλλά ήταν γεμάτη χαμόσπιτα. Και όταν ε, μετά ε, ρώτησα πόσα τέτοια χαμόσπιτα έχουν, μου είπαν 700.000 περίπου για μια χώρα που τότε είχε 3 εκατομμύρια κατοίκους. Ένα δηλαδή τέτοιο χαμόσπιτο είναι οικογένεια. Και γιατί? Γιατί κάθε εβδομάδα, κάθε οικογένεια έπρεπε να παρουσιάσει μια έκθεση για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το σπιτάκι της αυτό. Έτσι δημιουργείται ένα συγκεκριμένο πνεύμα ανάμεσα στον πληθυσμό, ο οποίος θεωρείται υποχρεωμένος να φροντίζει για τα σπιτάκια ας πούμε αυτά και έτσι να υιοθετεί μια συγκεκριμένη στάση με τον τρόπο αυτό το καθεστώς ήλεγχε όλο τον πληθυσμό. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα όπως είπαμε, θέλουν να ελέγχουν πλήρως ε, τον άνθρωπο. Και η έκθεση, η παρουσίαση του συναδέλφου μας το καταδεικνύει αυτό. Πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ακόμα σήμερα και θα τις έχουμε και στο μέλλον. Πρέπει να πάψει η ατιμορρησία στην Κορέα, αλλά ένας από τους ακτιβιστές, μάλλον ένας από τους προσκεκλημένους μας, είπε ότι η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα είναι τραγική. Χαίρομαι πάντως που η αντιπροσωπεία μας μπόρεσε να πάει στη χώρα αυτή. Ακόμα και αν τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε είναι τρομερά, παρόλα αυτά υπάρχει μια χτίδα φωτός. Έτσι ώστε στο μέλλον να μπορούμε να ελπίσουμε ότι ο πληθυσμός θα έχει πρόσβαση σε μια πιο αξιοπρεπή ζωή. Έχω εδώ στο μυαλό μου όλους τους κατοίκους και τα άτομα με αναπηρία που ίσως να μην έχουν καν το δικαίωμα στη ζωή στη χώρα αυτή. Και όπως έλεγα και νωρίτερα, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν δέχονται ε, τους ανάπηρους οι ανάπηροι δεν έχουν θέση μέσα σε μια τέτοια κοινωνία. Γιατί κάνουν το καθεστώς να ντρέπεται γι' αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι μιλήσαμε αρκετά για τα θέματα αυτά. Έτσι κι αλλιώς και στις επόμενες συνεδριάσεις θα έχουμε και άλλους προσκεκλημένους για να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά. Και θα έχουμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με τη Βόρεια Κορέα ξανά και ξανά. Και περνάω στο επόμενο σημείο. Πρόκειται για πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουινέα Κόνακρη. Ε, <coughs> λοιπόν, θα θυμόσαστε ίσως ότι το 2008 έγινε στρατιωτικό πραξικόπημα στην Γουινέα Κόνακρη. 156 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2009 και έλαβαν χώρα και μαζικές, μαζικοί μάλλον βιασμοί γυναικών και κοριτσιών στη χώρα από τις δυνάμεις ασφαλείας. Μετά είχαμε την εκλογική διαδικασία και πέρυσι έγιναν αυτές οι εκλογές. Ο κύριος Λάμστορφ ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας που πήγε για να παρατηρήσει τις εκλογές και ο οποίος δυστυχώς σήμερα δεν είναι εδώ γιατί συμμετέχει και αυτό στη συνεδρίαση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Είχαμε την έκθεσή του όμως, στην οποία υπογραμμίζει ότι οι αρχές της Γουινέας Κόνακρη πρέπει να έχουν ως στόχο ένα σύστημα δικαίου, ένα δημοκρατικό σύστημα. Οι εκλογές που θα γίνουν, έλεγε στην έκθεσή του, αποτελούν μια δοκιμή για την κυβέρνηση. Τον Δεκέμβριο θα γίνουν οι εκλογές και η κατάσταση είναι πάρα πολύ τεταμένη. Έχουμε εδώ τον Διευθυντή για την Αφρική από την Διεθνή Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος πήγε πέρυσι στο Κόνεκριν, ο κύριος Φλόρεντ Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα επικεντρωθώ στην παρέμβασή μου κυρίως στο θέμα της καταπολέμησης της ατιμορρησίας για ε, τη δημιουργία επίσης κράτους δικαίου. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ευκαιρία που μου δίνετε να μεταφέρω εδώ τη φωνή των θυμάτων μετά κυρίως το σφαγιασμό της 28 Σεπτεμβρίου 2009 στο στάδιο ε, της ε, και να μιλήσουμε για τις προσπάθειες που γίνονται για το κράτος δικαίου. Υπάρχει ο κύριος, ε, μάλλον ένα μήνα μετά από την ημερομηνία αυτής σφαγιασμού με ε, πληγές οι οποίες μολύνθηκαν. Στο τέλος, το θύμα, 37χρονος ε, αυτός ο οποίος μας εμπνέει σήμερα, έχασε τη μάχη με τη ζωή. Στις 28 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, στρατιωτικοί και παραστρατιωτικοί μπήκανε στο στάδιο της πόλης, δολοφόνησαν 156 ε, ανθρώπους και βίασαν 109 τουλάχιστον γυναίκες και κορίτσια. Στη συνέχεια, η ΦΙΔΕΑ που είναι μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, Γουινέα, Επίσης την προσοχή μας στο γεγονός ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη στα εκατοντάδες αυτά θύματα των σφαγιασμών και ότι οι κύριοι υπεύθυνοι εξακολουθούν να κατέχουν αξιώματα στη χώρα. Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας ήταν ε, άμεση. Οδήγησε σε πολιτική κρίση στην Γουινέα και η ίδια αυτή δράση μπορεί να βοηθήσει τώρα την Γουινέα να ολοκληρώσει την μεταπολίτευσή της, να περάσει δηλαδή σε ένα καθεστώς με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία θα αποκαταστούσε τα θύματα της 28 ε, Σεπτεμβρίου. Η Διεθνής ε, λοιπόν, Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με άλλες οργανώσεις αποφάσισε να στηρίξει δικαστικά τα θύματα της 28 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για 200 άτομα τα οποία συνοδεύουμε εμείς και βοηθάμε προκειμένου κάποια μέρα να υπάρξει δίκη. Βέβαια, πηγαίνουμε σημειωτών και εννοείται ότι τα εγκλήματα έχουν μείνει χωρίς να υπάρχει κανένας υπεύθυνο. Πέρα όμως από την καταπολέμηση της ατιμορρησίας που δεν πρέπει να μείνει μόνο στα λόγια, οι οργανώσεις μας στηρίζουν τα θύματα με την πεποίθηση ότι οι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις της σοβαρές ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αυτοί που εμποδίζουν την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στη χώρα και εξαιτία των θέσεων που κατέχουν φροντίζουν για την ατιμορρησία τους και βάζουν τα θύματα στην πάντα. Εμείς όμως θέλουμε να σπάσουμε αυτό το μπούμερανγκ της ατιμορρησίας. Το πρώτο εξάμεινο του 2012 θα υπάρξουν κοινοβουλευτικέ εκλογές που αποτελούν ένα επιπλέον σημαντικό βήμα για τον δημοκρατισμό στην Γουινέα. Η FIDH μέσω των δυνάμεών της έχει εντοπίσει το θέμα υπεύθυνων, να βρεθούν δηλαδή υπεύθυνοι για τα εγκλήματα της 28 Σεπτεμβρίου σαν ένα πολύ βασικό θέμα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να παραμένει ατιμορρησία. Είναι μεγάλη πρόκληση για τη νέα εξουσία, όπως ήταν και για την Σενεγάλη, ε, που έπρεπε να δικάσει τον ε, τέος ηγέτη του Τσάτ, το Σενεγαρέ. Η διεθνής ε, κοινότητα, λοιπόν, αναρωτιέται και οι οργανώσεις μας βάζουν αυτό το στίχημα. Δηλαδή, θέλουν να διαπιστώσουν ότι υπάρχει η θέληση και η δυνατότητα των αρχών να καταδικάσουν τους υπεύθυνους για τα εγκλήματα αυτά, να τους δικάσουν και να τους καταδικάσουν. Γιατί αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι τότε θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε νέα δράματα, τα οποία πάλι θα περιόριζαν τη φωνή των ε, θυμάτων. Αν όμως αποτύχουν, δεν θα κερδίσουμε. Το Διεθνές Δικαστήριο λοιπόν πρέπει να αναμειχθεί και να του δοθεί η ευκαιρία να δικάσει και να καταδικάσει τους υπευθύνους. Και εσείς λοιπόν με τη δικιά σας φωνή μπορείτε να απευθυνθείτε και στους διεθνείς εταίρους αλλά και στο καθεστώς της Γινέας για να σταματήσει αυτή η σιωπή, για να φανεί η δημοκρατία η οποία χρειάζεται, είναι αναγκαία για να φανεί η αλήθεια, να υπάρξει δικαιοσύνη και στη συνέχεια συμφιλίωση. Συμφιλίωση που, που δηλώνει ότι τη θέλει ο πρόεδρος Αλφακοντά και αποτελεί και ανάγκη. Δεν μπορεί να θυσιαστεί και συνοδεύεται από μια ελευθέρωση του λόγου αλλά και από εγγύσεις ότι σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες καταφεύγουν όλα τα καθεστώτα δεν θα επαναληφθούν. Ορίστηκε μία επιτροπή με... αλλά χρειάζεται μια πιο συγκεκριμένη εντολή και με τεχνική αρρωγή και πολιτική αρρωγή μπορούμε να φροντίσουμε η διαδικασία της συμφιλίωσης να γίνει μια διαδικασία αλήθεια δικαιοσύνη και στο τέλο της διαδικασία αυτής να έχουμε τη συμφιλίωση. Γιατί για να μπορέσουμε να γυρίσουμε τη σελίδα πρέπει να μπορέσουμε να την έχουμε διαβάσει ολόκληρη. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές ζητάμε από εσά να ενώσετε τις δικές σας προσπάθειες με εκείνες της Επιτροπής και των οργανώσεων που δρούν στην Γουινέα και να στηρίξετε τα θύματα για να μπορέσουν να φτιάξουν αυτό το κράτος δικαίου στην Γουινέα. Ορισμένα θύματα, χάρη στο πρόγραμμα που στηρίζομαι, θα μπορέσουν να έρθουν στις Βρυξέλλες και να πάνε και στη Χάγη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ώστε να εξηγήσουν τις δικές τους προσδοκίες. Χρειάζονται τη δικιά σας τη στήριξη, ατομική, συλλογική, έτσι ώστε να περάσουν από αυτό το στάδιο της μεταπολίτευσης και να προχωρήσουν ακόμα παραπέρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ό,τι ερωτήσεις έχετε είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω για λεπτομέρειες, ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική διαδικασία, τη συμφιλίωση κτλ. Η πολιτική διαδικασία είναι κάτι που έχει τεράστια σημασία σήμερα στη Γουινέα. Παραμένει κάτι το ασταθές υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που είναι τα διάφορα έθνη που αποτελούν την κοινωνία στην ε, Γουινέα. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να συμφιλιώσουμε τις κοινότητες μεταξύ τους, αλλά να συμφιλιώσουμε πάνω απ' όλα το κράτος με τον πολίτη. Που είναι μια πολύ βασική παράμετρος για την συμφιλίωση στη χώρα. Σας ευχαριστώ. <coughs> Ευχαριστώ. Ε, δεν ξέρω αν θέλει κάποιο το λόγο. Ο κύριο Φιλίπ Παντάμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να πάρω το λόγο. Άκουσα την ανάλυση του FIDL και συμφωνώ. Ε, φυσικά και εμείς θέλουμε ένα πρόγραμμα στήριξης της δικαιοσύνης, στήριξης των θυμάτων της 28 Σεπτεμβρίου και των γεγονότων που προηγήθηκαν. Και πιστεύω και εγώ ότι είναι ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάνει έκκληση στις αρχές, ώστε οι ανακρίσει των γεγονότων του 28 Σεπτεμβρίου να συνεχιστούν. Έχω να προσθέσω όμως δύο πράγματα. Πρώτον, είναι σαφές ότι το κράτος δικαίου είναι ο στόχος της δράσης της Ένωση στην Γουινέα. Και πέρα από την στήριξή μας στο FIDH, έχουμε και πρόγραμμα στήριξη στη δικαιοσύνη ευρύτερο και στήριξη των τομέων της δίκησης που συνοδεύουν δικαιοσύνη, γιατί κατά το παρελθόν ένα πρόβλημα που υπήρχε ήταν ο στρατός, ο οποίος δεν πειθαρχούσε. Δεν υπάκουε. Δεύτερον, για αυτή την υπόθεση, που είναι πολύ ευαίσθητη και λεπτή, προτιμήσαμε μια διακριτική διπλωματία, για την προσωπή δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε δηλαδή ότι η δουλειά που γίνεται και από το FIDH γίνεται πιο αποτελεσματικά αν γίνεται διακριτικά. Δηλαδή, πιέζουμε διπλωματικά αλλά διακριτικά και όχι ανοιχτά. Γνωρίζοντας ότι μιλάω για μας, έτσι δεν μιλάω για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μιλάω για τη δικιά μας, το δικό μας το ρόλο. Αλλιώς θα δημιουργούσαμε μια δυσάρεστη κατάσταση και μια αντίδραση αρνητική από την πλευρά της Γουινέας που θα δυσκόλευε τους στόχους μας. Το FTIH είναι σε επαφές με το ποινικό δικαστήριο που και αυτό παρακολουθεί την κατάσταση επιτόπου βρίσκονταν στη Γουνέ πριν από τρεις εβδομάδες νομίζω, ακριβώς για να εκτιμήσουν και αυτή την κατάσταση. Άρα υπάρχει κάποια πρόοδος όσον αφορά τις έρευνες που γίνονται για τα εγκλήματα. Αλλά μέσα στο 2012 θα φτάσει η ώρα της αλήθειας. Δηλαδή η δικαιοσύνη της χώρας είναι σε θέση ναι ή όχι να κάνει τις έρευνές της και τις ανακρίσεις της σε βάθος μέχρι να φτάσει στους υπεύθυνους οι οποίοι όπως ακούσαμε εξακολουθούν να κατέχουν αξιώματα στην ε, κυβέρνηση. Συνεπώς, η FIDH πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά της και το ποινικό δικαστήριο από τη δικιά του την πλευρά πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις ώστε ενδεχομένω να αποφασίσει κατά πόσο πρέπει ή όχι να ξανασχοληθεί με, την, ε, με τις έρευνες εκείνο εφόσον δεν ε, ε, υπάρξει πραγματική βούληση από πλευρά των αρχών στη χώρα. Ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε κύριε Βαντάμου. Υπάρχει κάποιος που να θέλει το λόγο. Δύο χρόνια μετά την σφαγή και περίπου ένα χρόνο πριν τις εκλογές κατάφερε ο πρόεδρος να βελτιώσει την κατάσταση στην ε, Γουινέα, αν και δεν πέτυχε πάρα πολλά. Τα πρώτα βήματα έγιναν. Βέβαια, τώρα η υπεύθυνοι της σφαγής θα πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Πρέπει να υπάρξει απονομή δικαιοσύνης. έτσι ώστε να μπορεί στη χώρα αυτή να υπάρξει και μια ελεύθερη πολιτική συζήτηση η Επιτροπή μας συμμερίζεται το γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αλλάξει η κατάσταση στη χώρα μετά τα όσα έγιναν το 2009. Και θεωρώ ότι και, το, και στο μέλλον θα ασχοληθούμε εντατικά με το δέρμα αυτό. Ο κύριος Παντάμι θέλει και πάλι το λόγο, νομίζω. Παρακαλώ. Merci, en fait. Euh, σας ευχαριστώ. Για να επανέλθω λίγο στα συμπεράσματά σας, θέλω να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, τα άτομα τα οποία αναφέρονται στη διεθνή έκθεση που ακολούθησε την σφαγή της 28 Σεπτεμβρίου και που είναι άτομα τα οποία κυκλοφορούν πάντα στο καθεστώς, εμπίπτουν στις ατομικές κυρώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά δεν υπάρχει συνεργασία. Είναι άτομα δηλαδή που βρίσκονται σε θέσεις, σε αξιώματα ισχύω και που δεν συνεργάζονται. Παρά τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην αναγνωρίζει τα άτομα αυτά στις θέσεις που βρίσκονται. Δεύτερον, από ό,τι κατάλαβα, υπογραμμίσατε την αργή διαδικασία, την έλλειψη εξελίξεων. Πρέπει όμως να επιμείνω και να σας πω ότι από τότε που ανέλαβε ο πρόεδρος Αλφακοντέ, ακόμα και αν μερικές φορές γίνονται λάθη, υπάρχει η βούληση να μπούμε σε ένα δίκαιο. Είδαμε ότι έγιναν διάφορα 3 ε, Απριλίου αλλά και το Σεπτέμβριο, 27 Σεπτεμβρίου, ο στρατός έμεινε ε, μακριά. Δεν κινητοποιήθηκε. Τα γεγονότα καταδικάστηκαν και η δυσκολία ήταν πολύ λιγότερη από ό,τι κατά το παρελθόν. Πιστεύουμε δηλαδή παρόλα αυτά ότι υπάρχουν κάπως θετικέ εξελίξεις όσον αφορά την ευαισθητοποίηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και τον ε, κύριο Ζέλ, ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Ερχόμαστε στο τέλος της ε, συνεδριασής μας κλείνουμε το σημείο αυτό που αφορά την Γουινέα Κόνακρη. Σήμερα κάναμε πραγματικά συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων, ε, διαφορετικών μεν, αλλά και ομοίων σε έναν βαθμό. Νότιο-Ανατολική Ασία, Δυτική Παππούα, Βερμανία, Αίγυπτο, Σουαζιλάνδη, Βόρειος Κορέα, ε, Γουινέα Κόνακρη. Συζητήσαμε για όλα αυτά τα θέματα. Παντού μιλούσαμε για το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον περιορισμό των ελευθεριών. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε την ε, εντύπωση ότι έχουν υπάρξει, με ξέρεις στη Βόρεια Κορέα, κάποιες αλλαγές, κάποια βελτίωση, κάποια βήματα προς τα εμπρός. Και αυτό είναι σημαντικό. Δημιουργείται έτσι η εντύπωση ότι σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν τώρα αρχίζουν σιγά σιγά τα πράγματα και βελτιώνονται. Αυτοί που έχουν κάνει τις παραβιάσεις, έχουν κάνει οι δεχθείς πράξεις, κατονομάζονται. Βλέπουμε λοιπόν πόσο κοινά είναι μερικά θέματα, παρόλο που μπορεί να βρίσκονται σε τελείως διαφορετικά σημεία του κόσμου. Ευχαριστώ όλους λοιπόν. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Ευχαριστώ την Γραμματεία για την προετοιμασία. Ευχαριστώ και την κυρία Γκόμες που έμεινε εδώ στρατιώτης πιστός μέχρι το τέλος. Είχαμε κάποια τεχνικά προβληματάκια. Ε, συμβαίνουν αυτά. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Καλό σα βράδυ.